Välkomna! Καλώς ήρθατε. Ας αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Καλώς ήρθατε. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Αυτό είναι το πρώτο σημείο μας. Μία αλλαγή θέλω να σας προτείνω για αύριο, για τις ψηφοφορίες θα θέλαμε τα θέματα της ε, κυρίας Ζαν ε, Λάμπερτ και του κυρίου Γιάν Κρέμερ το θέμα μάλλον, ε, η ενεργητική ένταξη και το θέμα 19 συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. Θα αρχίσουμε με αυτά την ψηφοφορία και θα συνεχίσουμε κανονικά. Δηλαδή θα αρχίσουμε με τα 16, 19 και 20. Θα έχεις ωραία. Πρακτικά τη συνεδρι... που έγινε στις 2 Μαρτίου, σας τα έχουμε στείλει, έχετε το λόγο αν θέλετε, μπορούμε να τα εγκρίνουμε πολύ ωραία. Okay. Eh, jag har två Έχω και δύο ανακοινώσεις. Υπάρχει web streaming σήμερα, να μεταδίδεται η συνεδρίαση δηλαδή στο διαδίκτυο, όπως και την προηγούμενη συνεδρίασή μας. Και... Υπάρχει ένας φάκελος για τις αντιπροσωπείες για την 5η Μαρτίου. Τα έχετε στα αγγλικά μέσα στο φακελό σας. Τα προσθέτουμε λοιπόν στα πρακτικά και περνάμε στον προϋπολογισμό 2010. Έχουμε τον εισηγητή, τον κ. Λάσλου Σούρεν. Κύριε Σόργεν Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Λάσλο Σέργεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή η σύνομη συνάντησή μαζί σας είναι τμήμα μια σειρά ε, όπου ως εισηγητής εγώ ε, κατά κάποιο τρόπο χτυπάω τη θύρα των ε, ειδικευμένων επιτροπών όπως το έκανε πέρσι η κυρία Χάουκ που ήταν τότε η συγκήτρια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό νομίζω. Γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία με τις ειδικευμένες επιτροπέ. Εσείς πολλά ξέρετε για το τι λείπει από το σχέδιο αυτό του προπολογισμού και γι' αυτό ενδιαφερόμαστε για να αποφασίσουμε στα σημαντικά πράγματα, να ακούσουμε τις απόψεις για να ξέρουμε πού θα ε, προβλέψουμε ε, τα εν λόγω κονδύλια. Από πέρσι επίσης είδαμε ότι από καιρούς καιρών ο εισηγητής για τον προεπολογισμό συνεργάζεται με συζητητές των ειδικευμένων ε, επιτροπών για τον προπολογισμό τους. Αυτό έγινε και τον Γενάρη φέτος πρώτη φορά και θα ξαναγίνει. Βέβαια κάποιοι συνάδελφοι θα φύγουν με τις εκλογές, πρέπει να αντικατασταθούν για το δεύτερο τμήμα του έτους από άλλους. Το δεύτερο τμήμα του έτους όμως θα είναι πάρα πολύ φορτωμένο με εργασία, γι' αυτό είπαμε ότι είναι καλό να δημιουργηθούν οι σύνδεσμοι από τώρα. Το πρώτο καινούργιο πράγμα φέτος ήταν οι κατευθύνες γραμμές για το σύνολο του προβολισμού. Ξέρετε ότι αυτό συζητήθηκε και ψηφίστηκε στην πρώτη σύνοδο του Μαρτίου. Αυτό είναι ένα νέο στοιχείο. Γιατί τα περασμένα έτη συζητιέται μόνο την Ολομέλεια του Απριλίου, λίγες μέρες πριν από την παρουσίαση του σχεδίου. Και βέβαια, είναι κάπως γελίο να μιλάμε για τις οι ιδέες μας και τα οράματά μας για το προσχέδιο του προπολογισμού δύο μέρες πριν υποβληθεί από την Κομισιόν. Τώρα έχουμε όμως πάνω από ένα μήνα και αυτό είναι πιο λογικό. Από την υψηλή ταχύτητα της διαδικασίας, συνήθιστα υψηλή ταχύτητα θα έλεγα, προέρχονται πολλά προβλήματα. Η ειδική επιτροφή είναι κατά κάποιο τρόπο θύμα της ταχύτητας αυτής, γιατί η προθεσμία για τις τροπολογίες ήταν 16 Φεβρουαρίου. Εγώ πήρα μια επιστολή από τον διακεκριμένο σας πρόεδρο εν ονόματι της Επιτροπής σας με τα πιο σημαντικά σημεία για τη δική σας επιτροπή όσον αφορά τον προπολογισμό του επόμενου έτους. Όπως είπα, ήταν μετά βέβαια τη λήξη προθεσμίας. Όταν διάβασα την επιστολή αυτή, ήμουνα μα ικανοποιημένο, γιατί σύμφωνα με τι δικέ μα εξημίσει, ίσω δεν ήταν σωστέ αυτέ, αλλά η δική μου εκτίμηση ήταν ότι το μήνυμα της επιστολής σας με τα τέσσερα αυτά σημεία έχει συμπεριληφθεί στο κείμενο. Ο πρόεδρος είπε ότι είναι απογοητευμένος που δεν αντικατοπτρίζουμε στη ε, επιστολή αυτή. Εγώ νομίζω όμως ότι αντικατοπτρίστηκε. Δεύτερον, εγώ ως εισηγητής θα μπορούσα να εντάξω το κείμενο αυτό στο δικό μας κείμενο. Όμως πρόεδρε, χωρίς να είμαι αντίθετος με το περιεχόμενο του μηνύματός σας, εγώ δεν θέλω να είμαι αντίθετος προς τους κανόνες και γι' αυτό περιόρισα το εύρος των κατευθυντηρίων γραμμών. Οι επιστολέ βέβαια μετράνε θεωρητικά τουλάχιστον, αλλά έχω ένα περιορισμό χρόνου. Και σύμφωνα με τη δική μου εκτίμηση και την ανάγκη της εναρμόνισης δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω την ίδια διατύπωση που υπάρχει στην επιστολή. Δεν θέλω όμως να διευκρινίσω τώρα ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Θα πρέπει πραγματικά να αναλάβουμε επίσημη δέσμευση στην πρώτη κατεύθυνση αυτή. Γιατί αυτή, η κρίση έχει μια κοινωνική διάσταση. Και εάν ενδιαφερόμαστε να στείλουμε ε, το σωστό μήνυμα στους Ευρωπαίους, το μήνυμα αυτό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της και ιδίως στο Κοινοβούλιο έχει αναλάγει τη δέσμευση να βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων. Θέλω να δώσουμε περισσότερη ασφάλεια στους Ευρωπαίους πολίτες, γιατί βρίσκονται σε μια ανασφαλή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουν τι θα γίνει με τα χρήματά τους ή με τις θέσεις εργασίας τους. Εάν λοιπόν μπορούμε κάτι να κάνουμε με τις περιορισμένες μας δυνατότητες, θα πρέπει να το κάνουμε και οι δυνατότητες μας είναι και τόσο περιορισμένες. Αν έχουμε κατά νου λοιπόν συμπληρωματικά κονδύλια βέβαια, <clears throat> είδατε τι γίνεται με το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης που αυτή τη στιγμή είναι γύρω να πάμε στο ευρωπαϊκό, πούμε, έχουμε ένα σχέδιο ανάκαμψη για πέντε δις για να λύσουμε αμέσως τα προβλήματα, αλλά αμέσως σημαίνει ότι σε λίγα χρόνια θα βάλουμε, θα θάβουμε το διοξείδιο του άνθρακα μέσα στην γη. Ε, δεν μπορούμε να ζητάμε από τον φορολογούμενο χρήματα για κάτι τέτοιο. Γι' αυτό ο εισηγητής σας προσπαθεί να έχει πιο αυστηρό αυστηρούς στόχους. Αναλύουμε δηλαδή πώς στο παρελθόν δαπανούνται τα διάφορα κονδύλια. Τι έχει γίνει δηλαδή όσον αφορά την εφαρμογή των προγραμμάτων. Αυτά τα κονδύλια που σωστά εφαρμόζονται μπορούν ίσως να αυξηθούν. Αλλά εκείνες οι γραμμές του προπολογισμού που δεν χρησιμοποιούν υπαρκώς, όχι μόνο σε ένα, αλλά σε περισσότερο το ενός έτη, θα πρέπει να δούμε ποια, ποιες είναι οι επιπτώσεις. Σε αυτό το θέμα, ο εισηγητής περιμένει τις κατευθείαν γραμμές των ειδικευμένων επιτροπών. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι για σας τα κονδύλια, οι γραμμές του προπολογισμού σας χρησιμοποιούνται επαρκώ. Εάν δεν χρησιμοποιούνται όμως επαρκώς, εμείς στην Επιτροπή Προπολογισμών δεν μπορούμε να λύσουμε γιατί δεν εφαρμόζονται ως πρέπει. Εσείς μπορείτε να το κάνετε. Υπάρχουν ίσως δικαιολογίες, αιτιολογήσεις. και θα πρέπει γι' αυτό εμείς στην αξιολόγησή μας να διακρίνουμε αν είναι δικαιολογημένη η υποχρησιμοποίηση αυτή ή όχι. Δεν θέλω να μακρηγορήσω πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφέρω απλώ ότι εν τω μεταξύ ετοιμάζουμε το δεύτερο μας έγγραφο εργασίας το οποίο θα υποβληθεί σήμερα και θα συζητηθεί στην Επιτροπή Προπολογισμών και θα υπάρχει μετά εδώ σε ένα παράρτημα όπου προσπαθούμε να δούμε ποια είναι τα κονδύλια που αρμόζουν σε αυτό το πρόγραμμα και δίνουν περισσότερη ασφάλεια στους πολίτες. Θα δώσω το έγγραφο εργασία αυτό στον δικό σας συζητητή του θέματος και θα θέλω να ξέρω κατά πόσο σύμφωνα με τη δική σας αξιολόγηση θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και άλλα κονδύλια εδώ. Γιατί εγώ θέλω αυτή η γραμμή των κονδυλίων να χρησιμοποιηθεί για την ε, βελτίωση του προπολογισμού το φθηνότερο. Ευχαριστώ να ακούσω τώρα τις ε, συμβουλές σας και τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστούμε. Για όσους δεν το γνωρίζουν, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στις 10 Φεβρουαρίου στη συνεδρίαση των συντονιστών αποφασίσαμε ότι θα συνέτασα εγώ μία επιστολή προς τον πρόεδρο της Επιτροπής λόγω του ότι άλλαξε η κατάσταση από οικονομικής πλευράς Ε, βιώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πλήττει με ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση και την αγορά εργασίας ε, όπως γνωρίζετε. Επίσης, ε, από πλευράς του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Κατάσταση υπάρχουν επιπρόσθετες πρωτοβουλίες και όχι μόνο για αυτό, αλλά για την καταπολέμηση της ένδυας και την γεφύρωση του χάσματος ε, του εισοδήματος ανάμεσα στις διάφορες ε, πληθυσμιακές ομάδες. Οπότε θελήσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτό τον τρόπο, την κατάσταση όπως ε, διαμορφώθηκε. Δεν έχει αλλάξει αυτό βέβαια, ακόμη βιώνουμε την ίδια κρίση και οι συντονιστές αποφάσισαν, πήραν αυτή την απόφαση για την επιστολή και αυτό κάναμε. Ο κύριος Ρή, ο εισηγητής μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτό είναι ένα ειδικό, μια ειδική χρονιά, η χρονιά, η χρονιά των ευρωεκλογών, κάτι το οποίο περιπλέκει το κανονικό μας χρονοδιάγραμμα. Ίσως όμως θα άξιζε να πούμε ορισμένα ε, λόγια για το πώς θα πρέπει να προωθήσουμε την εργασία μας. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι θα πρέπει να εργαστούμε με μεγάλη πίεση, με υψηλή ταχύτητα και επίσης να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι εξαιτία της προεκλογικής περίοδου μετά από την οποία μερικοί θα αποχωρήσουν, άλλοι θα παραμείνουν, θα επέλθουν αλλαγές. Σίγουρα ειδικά ως προς τα μέλη της Επιτροπής αυτής. Αυτή είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία εκείνων που προετοιμάζουν τον προϋπολογισμό, δηλαδή να εργαστούν το ταχύτερο δυνατό. Γι' αυτό απεστάλλει και αυτή η επιστολή από τον Πρόεδρο. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις προτεραιότητες που και εγώ έχω ε, υποβάλει γραπτός. Νομίζω ότι οι Σκιώδης, θα πρέπει να συναντηθούν την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου στο Στρασβούργο έτσι ώστε να αποφασίσουν για τις διάφορες προτεραιότητες. Νομίζω ότι υπάρχει σύμπτωση απόψεων. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, τότε μέχρι το τέλος της πρώτης συνόδου το Μάιο θα μπορέσουμε να υποβάλουμε το έγγραφο προς ε, μετάφραση και μέχρι τον ε, Αύγουστο 16-17 θα περιλάβουμε και τις τροποποιήσεις. Προτείνω λοιπόν προς τους συζητητές να συναντηθούμε στις αρχές Μαΐου να εργαστούμε εντατικά και να προσπαθήσουμε να εντάξουμε τις διάφορες υποδείξεις σε ένα έγγραφο το οποίο μετά θα υποβληθεί πριν από την προθεσμία. Ίσως θα ήταν σκόπιμο επίσης να υποβάλουμε ορισμένες ερωτήσεις στον κύριο Σούριαν, αλλά νομίζω ότι ήδη απάντησε. Από ό,τι κατάλαβα, θεωρεί ότι όλες οι ιδέες είναι ευπρόσδεκτες. Δεν έχω λάβει επίσημα τις υποδείξεις του, αλλά έχω δει το παράρτημα και ήδη έχω βρει ορισμένα σημεία όπου θα προβάλλουμε αντιρρήσεις. Θα ήθελα να πω όμως στον εισηγητή ότι θα θέλαμε να συνεργαστούμε μαζί του και οι πέντε προτεραιότητες που έχουμε υποβάλει και που απέστειλε ο πρόεδρος, τον κύριο Σούριαν, κάπως αργοπορημένα δυστυχώς, δείχνουν θα πρέπει να αντιδράσουμε κατά κάποιο τρόπο στην χρηματοπιστωτική αυτή κρίση, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα υπάρχει ε, απώλεια θέσεων εργασίας και αυτό και σε μία μεταβατική περίοδο. Θα πρέπει να ανακόψουμε αυτή τη διαδικασία, χρειάζονται χρήματα γι' αυτό και θα πρέπει να δημιουργήσουμε και νέες θέσεις εργασίας. Το θέμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Παγκοσμιοποίησης σχετίζεται άμεσα με αυτό το ζήτημα, είναι το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη και θεωρούμε ότι τα 500 εκατομμύρια θα πρέπει να αυξηθούν σε ένα δις, θεωρούμε ότι αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο. Το ίδιο ισχύει και για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, δηλαδή σημασία έχει να δαπανηθούν αυτά τα κονδύλια αποδοτικότερα για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και για να ανακόψουμε τα, τα διάφορα μειονεκτήματα που υπάρχουν στον κοινωνικό τομέα. Υπάρχουν ορισμένες αυξήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, κάτι το οποίο, συγγνώμη, μειώσεις, κάτι το οποίο όμως δεν είναι βάσιμο. Τώρα, ως προς την εκπαίδευση και την κατάρτιση, θεωρούμε ότι χρειάζονται περισσότερα κονδύλια σε αυτό το τομέα, διότι είναι βασική τομής της ε, μελλοντικής περίοδου που θα διανύσουμε, δηλαδή θα πρέπει να βρούμε νέους ε, τρόπους για την αντιμετώπιση της οικονομίας του μέλλοντος. Και τέλος, στις κατευθυντήριες γραμμές δεν βλέπουμε τι αντιμετώπιση υπάρχει για αυτούς που ζημιώνονται από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή για, τον, για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2010 θα πρέπει να εγγράψουμε κονδύλα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτό είναι αναπόφευκτο γιατί θα πρέπει να καταδείξουμε αλληλεγγύη προς τους ανθρώπους αυτούς Κάτι το οποίο είναι απόλυτα αναγκαίο στους, καιρούς, στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε. Αυτά προβλέπουμε και το γεγονός ότι ο πρόεδρος ε, προβάλλει αυτά τα ζήτηματα δείχνει ότι στην Επιτροπή υπάρχει συνένεση ως προς τα θέματα προτεραιότητας. Βεβαίως αυτό μπορεί να έχει διαφορετικές σταθμίσεις για τις διάφορες πολιτικές ομάδες, αλλά θα πρέπει να προωθήσουμε το όλο θέμα από κοινού. Και εάν ο συγητής της Επιτροπής Προϋπολογισμών δείξει ανοιχτό πνεύμα, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αυτά αρκούν επί του παρόντος, καθότι το έγγραφο εργασίας μόλις έχει συνταχθεί. Θα το εξετάσουμε και μέχρι τούδε δώσαμε προσοχή στα σημαντικότερα σημεία, στις προτεραιότητες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Κάλιονς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με τον κύριο Γιώργη. Είμαι αισιόδοξη ότι εν ώψη της ε, μεγάλης κρίσης που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι και πιο μεγάλη η πρόθεση συνεργασία μεταξύ των επιτροπών. Παρ' αυτά θα ήθελα να τονίσω το εξή. Και άλλα λεφτά και άλλα λεφτά και άλλα λεφτά. Το ξέρουμε τι συζήτηση ποια είναι. Αλλά θα είναι πολύ δύσκολο. Θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα συντονισμό των πόρων στους ε, τομεί που μα φαίνεται πάρα πολύ σημαντικοί. Δηλαδή κατά του κοινωνικού αποκλεισμού, υπέρ τη επαγγελματική ειδίκευση και δημιουργίας θέσεων απασχόληση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα νέα προγράμματα που θέλουμε τώρα να εισαγάγουμε με προγράμματα πιλότους, προγράμματα ε, παιδείας για τους ε, μαθητευόμενους παραδείγματος χάρη να αναπτυχθούν. Λυπούμε γιατί δημιούργησε την εντύπωση ότι ο εισηγητής αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη των συστημάτων ασφάλειας. Αυτό είναι ένα πράγμα γενικά η ασφάλεια στην Ευρώπη, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε το θέμα της κοινωνικής ασφάλισης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Στίβεν Χιούς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να συμφωνήσω με τη Σάρμπα. Ελπίζω ο εισηγητής ε, να μεταφέρει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών ε, το μήνυμα ότι όχι μόνο δεν ανταποκρίνθηκαν στις προσδοκίες μας αλλά και ε, κυρίως αυτοί που πλήττονται από την οικονομική κρίση ε, είχαν προσδοκίες ε, που δεν καλύπτονται. Αυτό ισχύει για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι συγκεκριμένο που πρέπει να δούμε στα πλαίσια των τροπολογιών είναι η ζωτική σημασία του να διατηρήσει ο κόσμος τη δουλειά του. Στη Στοκχόλμη πριν από λίγες εβδομάδες, εκεί που ήμασταν με το Γιάννη δηλαδή, Μάθαμε ότι για τους μεταλλορύχους θα υπάρχει 25% μείωση του χρόνου εργασίας, 20% ε, μάλλον μείωση του χρόνου εργασίας ε, και θα εφαρμοστεί αυτό το σύστημα που ονομάζεται Smart Working, ευφυής απασχόληση θα πρέπει να προβλεφθεί μια κοινοτική παρέμβαση όχι μόνο μέσα από το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση αλλά και μέσα από τα διαρθρωτικά ταμεία. Μόνο έτσι θα αποφύγουμε να χάσουν κάποιοι τη δουλειά τους γιατί συνέχεια θα μετεξελιχθούν σε μακροχρόνια άνεργους και θα μπορέσουν ε, έτσι να ξεπεράσουν την οικονομική κρίση αναπτύσσοντας και τις δεξιότητές τους. Νομίζω ότι ε, θα πρέπει να κάνουμε αυτές τις παρατηρήσεις μέσα στις τροπολογίες για τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων και όπως έλεγα και στην αρχή ελπίζω ο εισηγητής να περάσει το μήνυμα στην Επιτροπή Προϋπολογισμών για την οικονομική κρίση. Σας ευχαριστούμε. Δεν έχω κανέναν άλλον ομιλητή, απλά να προσθέσω κι εγώ, όπως ακούσαμε και από συναδέλφους, να τονίσουμε λοιπόν ότι υπήρχε πίεση για αυτή την επιστολή. Υπήρξε μεγάλη ομοθυμία ότι Δηλαδή ήταν, ε, παράξενο αν εμείς ε, δεν ε, καλύψουμε τις ανάγκες του πληθυσμού της Ευρώπης λόγω του, της οικονομικής κρίσης που πλήττει σε μεγάλο βαθμό την Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν με πολλούς και διάφορους τρόπους να την αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση ε, να μην αποκλείονται από την αγορά εργασίας ε, οι υπήκοοι της Ένωσας ε, και επίσης να είμαστε προετοιμασμένοι όταν υπάρξει ανάκαμψη. Δεν έχουμε πλήρως αξιοποιήσει τις δυνατότητες που έχουμε για την κατάρτιση ε, ορισμένοι ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει χρόνος. Τώρα έχουμε χρόνο και είναι σημαντικό να γίνει αυτό και με τη βραχυπρόθεσμη πρόπτικη και τη μακροπρόθεσμη πρόπτικη. Γι' αυτό κάνουμε αυτή την πρόταση από πλευρά σε κοινοβουλίο και την διαβάσαμε και στην Επιτροπή Προϋπολογισμού. Θα ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Σέργεν τώρα για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θέλω να, κλείσω, να κλείσω τη συζήτηση. Νομίζω ότι θα τη συνεχίσουμε και στο μέλλον θα ήθελα όμως να επαναλάβω ορισμένα όσα άκουσα. Στο, στην ιστοσελίδα κόπου μπορείτε να βρείτε το έγγραφο εργασίας μου και υπό τον τίτλο «Ασφάλεια για τους Ευρωπαίους πολίτες» το πρώτο σημείο είναι να απαντήσουμε στην οικονομική παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Άρα η ασφάλεια είναι η μεγάλη κάλυψη, η ομπρέλα αυτή και μετά μιλάμε για ασφάλεια εργασίας, δημιουργία θέσεων εργασίας, υποστήριξη θέσεων εργασίας και ε, στόχοι της Λισαβόνας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, Πρόεδρε, ότι όχι μόνο το Ταμείο Παγκοσμιοποίηση, εσείς νομίζω το είπατε αυτό, αλλά και η ίδια η πολιτική συνοχής και το Ταμείο Περιφερειακής Συνοχής είναι κεφαλαιόδου σημασίας εάν μιλήσουμε για την αύξηση ΑΕΠ και δημιουργία θέσεων εργασίας, τότε η κατάσταση θα ήταν καλύτερη. Δηλαδή μιλάμε για στοχοθετημένη χρήση των χρημάτων και όχι περισσότερα χρήματα. Θα πρέπει όμως να επηρεάσουμε στην καταβολή, στη δαπάνη των χρημάτων. Θα πρέπει να γίνει σωστή στοχοθέτηση. Διαφορετικά δεν μπορούμε να διαχειριστούμε αυτό το πλαίσιο. Μιλήσατε για το θέμα των πιλωτικών σχεδίων. Είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Νομίζω ότι είναι υποχρέωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αποστείλει τα πιλωτικά σχέδια, όχι λεπτομερώς, αλλά ως προς το βασικό περιεχόμενο στην Επιτροπή, πριν από το καλοκαίρι. Γιατί ε, το ζήτημα αυτό δεν αφορά την προεκλογική περίοδο. Αν υπάρχει ένα πιλωτικό σχέδιο ως Επιτροπή ή μονομένα μέλη, θα τα αποστείλω αυτά τα σχέδια στην Επιτροπή γιατί έτσι αυτά τα πιλωτικά ε, προγράμματα μπορούν να τύχουν διαχείρισης ε, αργότερα. Θα έχουμε την ε, επιστολή εκτελεσιμότητας και μετά θα αποφασίσουμε όταν θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό. Πρέπει να γίνει λοιπόν τώρα. Θα ήθελα να αναφέρω, όπως είπε και ένας άλλος συνάδελφος, ότι θα πρέπει να να έχουμε ένα δις στο Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Αλλά το πρώτο έτος λειτουργίας μόνο το 4%, λιγότερο από το 4% χρησιμοποιήθηκε, το δεύτερο χρόνο λιγότερο από 10%. Το 2009 δεν είναι εύκολο να προβλέψουμε, αλλά φαίνεται ότι αυξάνεται ε, η χρήση, αλλά πάνω από τα 500 εκατομμύρια. Μπορώ να δώσω μάχη για περισσότερα χρήματα, αλλά θα χάσουμε, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία και υπάρχει στις κατευθυντήριες γραμμές που υπέδειξα είναι ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τους ε, κανόνες του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης έτσι ώστε να είναι περισσότερο αποτελεσματικό. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί και όταν χρησιμοποιήσουμε όλα τα κονδύλια τότε μπορούμε να ε, αποζητήσουμε περισσότερα. Διαφορετικά θα πρέπει να θεωρήσετε ότι υπάρχουν δυσκολίες και στα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο δεν ήταν ποτέ πολύ γενναιόδωρο να δώσει χρήματα στο ταμείο αυτό. Κάνει μεγάλο λάθος βέβαια που αντιτίθεται σε αυτή την ιδέα των ε, περισσότερων χρημάτων. Αυτό είναι προβληματικό, άκρος προβληματικό. Τέλος, για να σας εξηγήσω το γεγονός ότι η δική μας συνεργασία ήταν πολύ καλή, θα ήθελα να τονίσω ότι αυτές οι κατευθυντήριες ε, γραμμές που ψηφίσατε στην Ομέλεια και σας ευχαριστώ γι' αυτό και εξαιτίας αυτής της ψηφοφορίας θα πρέπει να δούμε την χρηματοοικονομική κρίση και τις επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα στις θέσεις εργασίας, καλύτερη εφαρμογή διαρθρωτικών ταμείων και ούτω καθεξής. Αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει, ιδιαίτερα η κοινωνική συνοχή, πάλι αναφέρεται για να αποφύγουμε τον κίνδυνο απώλειας θέσεων εργασία, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και να βοηθήσουμε και το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Προσπαθήστε να βρείτε χρόνο για να διαβάσετε το έγγραφο εργασίας μας και θα δείτε τον ενδυνάμει κατάλογο των προτεραιοτήτων τις στοχοθετήσεις μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας και ελπίζω αυτή η συνεργασία να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για το μέλλον. Τέλος, υπάρχει μια προθεσμία υποβολή τροπολογιών στις 9 Σεπτεμβρίου μέχρι το 12 το μεσημέρι. Πολύ δύσκολη αυτή η εργασία. Τότε η Επιτροπή θα πρέπει να συνέλθει. Τα μέλη θα πρέπει να κάνουν την εργασία αυτή μία εβδομάδα πριν. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Ο καθένας θα ψάχνει για το πού βρίσκεται και δεν είναι ο κατάλληλος χρόνος, η κατάλληλη χρονική στιγμή. Θα πρέπει να υποβάλλετε τροπολογίες σε επίπεδο επιτροπής, κάτι το οποίο θα δώσει μια μεγάλη όθηση που ελπίζω να μπορέσουμε να διαχειριστούμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας φυσικά. Θα ήθελα απλά να σας ενημερώσω για το εξή. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό μέχρι στιγμής για διάφορους λόγους. γιατί υπάρχουν διάφορα κριτήρια και ε, είχε συσταθεί σε μια εντελώ διαφορετική κατάσταση που αυτή επιβιώνουμε σήμερα. Και γι' αυτό μιλάμε για, για αλλαγή της χρήσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την ε, παγκοσμιοποίηση στα πλαίσια των συζητήσεων που έγιναν. Όπως σας έλεγα προηγουμένως ότι συζητούμε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση σήμερα. Δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, να το επικαλεστούμε αν θέλετε ως επιχείρημα για την αυξημένη χρήση αυτού του Ευρωπαϊκού Ταμείου. Αυτό τοποθετείται στις, στα πλαίσια των συζητήσεων που κάνουμε γενικότερα για την αλλαγή της κατάστασης. Όχι, δεν μπορούμε να το τοποθετήσουμε μόνο στα πλαίσια του προπολογισμού δηλαδή. Λοιπόν, ευχαριστούμε που ήρθατε. Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία και λίγη αυτό το σημείο για σήμερα. Όπω σα έλεγα λοιπόν, τώρα θα ασχοληθούμε με την ίδια τροποποίηση του κανονισμού 1927 2006 για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Η κυρία Στάουνερ είναι η συγγήτριά μας. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Μετά από μια συνομιλία την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο με τους κοιόδης συγητές, υπέβαλα την πρόταση που βλέπετε στην, ε, στον κατάλογο ψηφοφορίας. Οι περισσότερες μου επιστροφολογίες ε, να αποσυρθούν, πράγμα που έγινε. Πάνω από 20 έχω αποσύρει τώρα και να συνεχίσουμε τη, να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας συγγνώμη, σε τρία-τέσσερα σημαντικά θέματα για να μπορέσουμε να τελειώσουμε γλίγορα. Αλλά νομίζω ότι υπήρχε συνένεση την περασμένη εβδομάδα στην συνομιλία αυτή που είχαμε γιατί θα πρέπει το ταμείο παγκοσμιοποίησης να χρησιμοποιηθεί κατά το δυνατόν καλύτερα και γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε κάποιες αλλαγές, να μην αναβάλουμε ΣΑΗ, e, αλλά να δράσουμε τώρα. Δεν μπορώ λοιπόν αυτή τη στιγμή παρά να σας πω ότι αυτή η γραμμή του να ακολουθήσουμε την πρόταση Κομισιόν χωρίς καμία τροποποίηση δεν μου φαίνεται ότι είναι λογική και εφαρμόσιμη. Θα πρέπει και ελπίζω να συμφωνήσετε πάνω σε αυτά. Καταρχήν, να έχουμε αυτό το 20% ακριβώς όπως το έχουμε στο ΕΣΕΦ θα ήθελα να σας υπενθυμίσω την έκθεση της συναδέλφου Γιάντς, όπου είχαμε και εμείς ως ομάδα συμφωνήσει. Και νομίζω αυτό το κατακοπή πρέπει να εισαχθεί και εδώ, στο ΕΖΕΦ. Νομίζω θα ήταν εύκολο εδώ. Και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να σας βρει σύμφωνους. Εγώ μπορώ να συμφωνήσω και θα πρέπει και εσείς να συμφωνήσετε. Αυτή είναι η τραπολογία 47. Το ίδιο θα ήθελα να κάνω, είχαμε πει, η ομοιομορφία αυτών των διαφόρων ταμείων. Τώρα, καλός, κακός, άλλο θέμα αυτό. Αλλά, εν τελευταία αναλύση, είναι αλληλένδετα τα δύο ταμεία αυτά ενίσχυσης και γι' αυτό όσον αφορά το ύψος της συγχρηματοδότηση να ε, προσανατολιστούμε στο Ταμείο ΡΣΕΦ Δηλαδή μπορώ να συμφωνήσω όπως είπα την Κομισιόν σε μια συγχρηματοδότηση 75% από την Κομισιόν όπως το θέλουν και ορισμένοι ε, συνάδελφοι απολύτως απαραίτητο. Αυτό νομίζω θα απλουστεύσει τα πράγματα και έτσι δεν θα χρειαστεί τα διαφορα κρατημένα να έχουν διαφορετικά ε, διαφορετικούς τρόπους ε, <clears throat> Θα ήθελα επίσης να συστήσω την ε, τροπολογία 43 τη Ανέλφου Σουρέτερ που μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Μπορώ να συμφωνήσω και με την τροπολογία 51 των φιλελευθέρων του συναδέλφου Κοτσιλόβο ή τέλο πάντων της φιλελεύθερης ομάδας ότι οι πόροι αυτοί θα πρέπει να δοθούν συμπληρωματικά στους εργαζόμενους επιπλέον δηλαδή από αυτό που χορηγείται Τώρα μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ λογικό και σημαντικό επίσης. Για να απομείνω αρκετά για τους εργαζόμενους. Επίσης συμφωνώ με τις τροπολογίες, υπάρχει και μια δική μου νομίζω, τέλος πάντων τις 45 και τις 35 της συναδέλφου Σρέντερ, να μην ε, προβλέπονται πόροι για τεχνική ενίσχυση από τη σκοπιά τη Κομισιόν, γιατί θέλουμε οι πόροι αυτοί να δοθούν πλήρω σε εκείνου που αναφέρονται στον τίτλο, δηλαδή στου εργαζόμενου. Και όχι να χρηματοδοτήσουμε κάποιες δραστηριότητε τη Κομισιόν με τα χρήματα αυτά. Αυτά σε γενικέ γραμμέ. Βλέπετε ότι εγώ περιόρισα την προσοχή μου σε τρία-τέσσερα σημαντικά σημεία και ελπίζω όλα τα μέλη της Επιτροπής μας να μπορέσουν να συμφωνήσουν με αυτά που προτείνω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Έχουμε διάφορες ομιλητές. Ο κύριος Ναρένιο Κομπάρ και ο κύριος Στίβεν Χιούς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εντάχει, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την εργασία της ε, Γκαμπρίελα Στάουνερ, της ε, εισηγήτριας, διότι κατά τις τελευταίες συζητήσεις και τις τροπολογίες έδειξε την ε, κατάλληλη πολιτική ευελιξία και ευφυΐα. Γι' αυτό αυτό θα ήθελα καταρχήν να αναφερθεί. Θα πρέπει να διευκρινίσω τα θέματα ουσίας από δικής μου πλευράς και θα ήθελα να πω ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, έκτακτη κατάσταση, γι' αυτό η Επιτροπή προτείνει την αλλαγή ενός μέσου κατά εξαιρετικό τρόπο. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να κρίνουμε ίσα άνισες ε, συνθήκες θα πρέπει να γίνει η μεταρρύθμιση αυτού του μέσου. Όχι μόνο από οικονομικής πλευράς αλλά και πολιτικής. Υπό αυτή την έννοια θα ήθελα να σας πω ότι το κείμενο της Επιτροπής ε, στο σύνολό του αποτελεί πολιτική απάντηση και νομίζω θα πρέπει να ε, αντικατοπτρίζεται η εμβέλεια αυτού του ζήτηματος και να έχουμε και ένα κατάλληλο μέσο, τροποποιημένο μέσο σε πρώτη ανάγνωση. Γιατί μου φαίνεται και καθίσταται σαφές ότι θα πρέπει να εγκρίνουμε αυτό το αίτημα που δεν είναι μόνο των πολιτών, διότι η, απερι... η ανεργία, με συγχωρείτε, είναι το πιο σκληρό πρόσωπο αυτής της χρηματοπιστωτικής κρίσης και εμείς θα πρέπει να δώσουμε μια πολιτική απάντηση. Είναι γεγονός ότι ίσως πέλθουν αλλαγές συζητήσιμες, αλλά νομίζω ότι διανύουμε μία κατάσταση όπου θα πρέπει να δώσουμε μία ταχύτατη, τάχιστη απάντηση προς τους πολίτες και γι' αυτό προτείνω το κείμενο της Επιτροπής να εγκριθεί ως έχει. Δεν συμφωνώ με εκείνους που θέλουν να διευρύνουν το κείμενο. Νομίζω ότι ούτε από πλευράς συσταλτικής ούτε διασταλτικής θα επέλθουν ουσιώδεις αλλαγές. Θα πρέπει να εγκρίνουμε λοιπόν την πρόταση της Επιτροπής εκτός και αν υπάρχει ένα συμβιβασμός ομάδων για να τροποποιήσουμε δύο-τρία σημεία χωρίς ε, να θίξουμε την ε, ουσία. Πρέπει να καταβληθεί πολιτική προσπάθεια υπέρ των πολιτών. Επίσης πιστεύω ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να πούμε στους πολίτες ότι δεν μπορούμε να τελειοποιήσουμε αυτό το ταμείο, δηλαδή να μην χρησιμοποιήσουμε ορισμένα κονδύλια που όπως είπε και η Γκαπριέλα είναι χρήματα τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί εδώ και δύο χρόνια. Πώς θα εξηγήσουμε στους πολίτες ότι ε, δεν θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα κονδύλια. Άρα η θέση μου είναι απλή, απλούστατη. Θα πρέπει να προωθήσουμε αυτό το κείμενο το ταχύτερο δυνατόν και κατά συνενετικό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χιούς έχει και μετά η κυρία Γιουκνα. Ο κύριος Χιούς. Ο συνάδελφος που ήταν σκιώδης δεν είναι παρόν, γι' αυτό θα ήθελα να πω ορισμένα λόγια. Δεν χρειάζεται να πω πολλά, διότι η θέση μας είναι σαφής εξ αρχής. Ο Ζαν Λουί δεν έχει υποβάλει τροπολογίες, διότι θα πρέπει να συμφωνηθεί αυτό το κείμενο, όπως είπε και ο κύριος Εσχομπάρ, το συντομότερο δυνατόν. Και δεν θα πρέπει να υπάρχει τροχοπέδι πιστεύω ότι οποιαδήποτε τροπολογία θα έθετε παγίδες στο Συμβούλιο. Θα πρέπει να επέλθει συμφωνία, ελπίζω την ε, Πέμπτη, δηλαδή να μην υποβάλουμε νέες τροπολογίες μέχρι την Πέμπτη έτσι ώστε να έχουμε ένα καθαρό ε, κείμενο. Η κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να ζητήσω από τις υπηρεσίες να κοιτάξουν την μετάφραση στα λιθουανικά, διότι υπάρχουν ορισμένα συντακτικά λάθη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ευέλικτη θέση της. Φαίνεται ότι θα είναι δύσκολο να επέλθει συμβασμός, αλλά βλέπω ότι ολοένα και περισσότεροι συνάδελφοι υποστηρίζουν την συνένεση, τη συνενετική αυτή διαδικασία και θέλουν να υποστηρίξουμε την θέση της Επιτροπής. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε τα βασικά ζητήματα τα οποία ανέφεραν ορισμένοι συνάδελφοι, δηλαδή τη σημασία του Ταμείου στην τρέχουσα κατάσταση. Αν δεν δώσουμε μία απάντηση, αν δεν ανταποκριθούμε, θα είναι δύσκολο να το εξηγήσουμε αυτό στους ψηφοφόρους μας και στους πολίτες που αναμένουν την υποστήριξη όχι μόνο από τις κυβερνήσεις αλλά και από το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την ταχύτατη αυτή διεκπαιρέωση, τον κύριο Στόμπι Γιάργενσον, τον οποίο συνάντησα ο οποίος μου ανέφερε ότι στα πλαίσια του Συμβουλίου οι διαπραγματεύσεις ήταν ιδιαίτερα επιτυχής και τα περισσότερα μέλη κατανοούν τη σημασία του Ταμείου. Γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε αυτή την εργασία τάχιστα για να ανταποκριθούμε στην τρέχουσα κατάσταση. Πιστεύω ότι οι άλλες διαφωνίες δεν είναι σημαντικές και δεν πρέπει να χάνουμε πολύτιμο χρόνο. Λυπάμαι κυρία Στάουνερ, δεν ήμουν σε θέση να συμμετάσχω στην συνάντηση των σκιωδών στο Στρασβούργο, αλλά από τα email κατανόησα ότι η πολιτική μου ομάδα θα υποστηρίξει το κείμενο της Επιτροπής και δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν οποιασδήποτε παρεξηγήσεις. Ε, μεταξύ φιλελευθέρων και δημοκρατών. Θα ήθελα και οι άλλες ομάδες να έχουν μια ευέλικτη άποψη για το Ταμείο Αντιμετώπισης της Παγκοσμιοποίησης και θα ήθελα να αντιδράσω στις ιδέες ε, το, του εισηγητή από την Επιτροπή Προπολογισμών που είπε ότι το Ταμείο Αντιμετώπισης Παγκοσμιοποίησης δεν χρησιμοποιήθηκε ε, πλήρως. Δεν έχει σημασία πόσα κονδύλια χρησιμοποιήθηκαν το πρώτο και το δεύτερο έτος. Σημασία έχει πώς χρησιμοποιήθηκαν και είμαι σίγουρη ότι χρησιμοποιήθηκαν σωστά αν αναλύσουμε την εφαρμογή από τα κράτη-μέλη και δούμε τα διάφορα παραδείγματα που καταδεικνύουν ότι υπάρχει αλληλεγγύη με τους πολίτες οι οποίοι βρέθηκαν εκτός αγοράς εργασίας. Σημασία έχει η αποτελεσματική χρήση του Ταμείου. Δεν έχει σημασία αν δεν χρησιμοποιείται, αν δεν έχει παρά μία βραδία πορεία, γιατί οι διαδικασίες είναι περίπλοκες και νομίζω ότι σύν το χρόνο θα το αποφύγουμε αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή και για την πρωτοβουλία της, όχι μόνο στα έγγραφα, αλλά σε αυτά που ανέφερε ο κύριος Γιόργενσεν, δηλαδή οι διαδικασίες θα κινηθούν παράλληλα έτσι ώστε να, να βραχύνουμε το χρόνο εφαρμογής και να επιταχύνουμε δηλαδή την εφαρμογή και να μην χάνουμε χρόνο. Από ό,τι κατάλαβα, μερικές φορές ε, αναβάλουμε τις αποφάσεις μας και τις αναθέτουμε σε άλλες ομάδες εργασίας. Θα πρέπει να ανταποκριθούμε εντάχει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπούσελ Μάθιος και ο κύριος Χάσε Φερέιρα. Φίλιπ, έχεις πρώτος το λόγο. Ευχαριστώ. Ε, τη σύντομη παρέμβασή μου θα την αρχίσω λέγοντας ότι συμφωνώ με τον συνάδελφο Ναράζο Έσκομπαρ. Δεν θέλουμε ε, ε, θέλουμε στην πρώτη ανάγνωση συμφωνία με συνένεση. Ε, κατά τη γνώμη μου αυτό δεν συνεπάγεται όμω ότι δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε, να κερδίσουμε υποστήριξη για κάποιε τροπολογίε, ε, για τι οποίε κανονικά θα υπήρχε ευρεία συμφωνία. Ο εισηγητή έχει αποσύρει τι περισσότερε τροπολογίε και έχει αποκρισταλώσει την άποψή του μέσα σε λίγε τροπολογίε με αυτό το στόχο, να καταλήξουμε συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Οπότε και εμεί μέσα από αυτή την οπτική γωνία πρέπει να το δούμε και ε, ο κ. Κοτσιλόβο από του ε, φιλελευθέρου ε, νομίζω θα συμφωνήσει μαζί μα, μπορεί να υποστηρίξει κάποιε από τι τροπολογίε μα. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε δυσκολίε ούτε να κολυσιοργούμε. Αυτό στο οποίο αποσκοπούμε είναι αυτή η συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση να μην παρακάμψει το Κοινοβούλιο επειδή η Επιτροπή και το Συμβούλιο ισχυρίζονται αυτό πρέπει να κάνουμε και άρα δεν χρειαζόμαστε το Κοινοβούλιο. Ε, αλλά να έχουμε κάποια σημεία επιτάπητο ε, τα οποία θα συζητηθούν. Εάν τελικά για αυτά τα σημεία δεν καταλήξουμε συμφωνία, κατά τη διάρκεια τη συζήτηση α απορροφηθούν από τη συζήτηση, τα εγκαταλείψουμε κατά τη διάρκεια τη συζήτηση. Αλλά συγγνώμη, να μην τοποθετηθούμε καθόλου εν ώψη αυτή τη συμφωνία. Ε, ε, δεν συμφωνούμε. Θέλουμε συνένεση, θέλουμε συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση, αλλά να τοποθετηθούμε κιόλα. Σα ευχαριστούμε. Ο κύριο Χάσε Φερέιρα και η κυρία Σρέτερ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να συγχαρώ την Γκαπριέλ Στάουνερ, την εισηγήτριά μας, για το 75%. Ε, υπέρ το οποίο ήμασταν κάποιοι από εμά κατά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ η κυρία Σρέντερ και ο κύριο Χέλμερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω ότι ε, την περασμένη εβδομάδα ε, είχαμε μία συμφωνία μεταξύ ε, σκιωδών εισηγητών και τελικά η κυρία Στάουνερ το αποτυπώνει αυτό μέσα στο έγγραφό τη. Μπορεί να υπάρξει μία αποτελεσματική χρήση του Ταμείου. Επικεντρώσαμε την προσοχή μας στα βασικά σημεία. Απέδωσε τη δέουσα σημασία η κυρία Στάουνερ σε αυτά τα σημεία και συμφωνεί η πολιτική μας ομάδα για το 75%. Γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι ότι Κανονικά στην Ολομέλεια θα ε, επιφέρουμε βελτιώσεις στο κείμενο, τόσο ώστε να υπάρχει και συμφωνία με το ΕΚΤ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και να λειτουργεί πιο εύρυθμα το σύστημα. Ε, πρέπει να διατηρηθεί οπωσδήποτε σχετική τροπολογία. Επ' αυτού είχαμε συμφωνήσει. Εξάλλου είχαμε πει ότι είναι απαραίτητη αυτή η τροπολογία στο βαθμό που ο στόχο είναι να ρυθμίσουμε τα προβλήματα στην Ολομέλεια, αλλά αντίθετα για το 75% εμεί κανένα πρόβλημα δεν έχουμε. Και για τις λοιπές ε, προτάσεις θα σας υποστηρίξουμε κυρία Στάουνερ και χαιρόμαστε πάρα πολύ που αποσύρατε κάποιες από τις τροπολογίες που ενδεχομένως θα είχαν δημιουργήσει προβλήματα. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι ε, με το στόχο να λειτουργήσει εύρυθμα το Ταμείο όλα όσα κάνατε ήταν πάρα πολύ χρήσιμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, ακούω τη συζήτηση και έχω λένε περισσότερο την εντύπωση ότι δεν είναι ρεαλιστική η συζήτηση οι πολίτες της Ένωσης περιμένουν να τους στηρίξουμε, ακούσαμε. Ακούσαμε ότι δεν καταλάβουν οι πολίτες άμα δεν ε, ε, ε, καλύψουμε τις προσδοκίες τους. Εμένα, κανένας από τους ψηφοφόρους μου δεν μου είπε ότι περιμένει τη δική μας βοήθεια. Κανείς δεν μου είπε ότι δεν θα καταλάβει αν εμείς δεν ανταποκριθούμε σωστά στην κρίση. Αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, ναι, έχει πολλά κονδύλια για ταμείο. Αλλά ε, αν το συγκρίνουμε με την ε, μεγάλη οικονομική κρίση ε, δεν είναι τίποτα, είναι ψίχουλα. Και αν σκεφτείτε και πόσα χρήματα δαπανούμε για τις κοινωνικές δραστηριότητες, για την ανεργία, για την κατάρτιση ε, και διάφορες ε, ενέσεις των που κάνουν κάποια κράτη-μέλη στις οικονομίες τους είναι ψίχουλα αυτά τα λεφτά του Ευρωπαϊκού Ταμείου και πραγματικά ε, για ποιους περνιόμαστε θα έλεγα που ασχολούμαστε με αυτά τα ψίχουλα και λέμε ότι, τα, ότι μας περιμένουν οι πολίτες της Ένωσης για να δουν τι θα κάνουμε αν δηλαδή σαν λευκοί υπότε θα έρθουμε να τους σώσουμε συγγνώμη έρθουμε στα στα συγκαλά μας. Ε, μιλάμε για ένα περιθωριακό ποσό έτσι, ε, ε, σε σχέση με την κλίμακα της κρίσης. Εμείς στη Σουηδία λέμε ότι περιμένουν πολλά στόματα να φάνε από την ίδια τροφή. Είναι αλήθεια ότι ε, έχουμε πολλές τρύπες να καλύψουμε με το Ευρωπαϊκό Ταμείο, αλλά είναι σημαντικέ όλε οι παρεμβάσει. Γιατί κάποιοι άνθρωποι τα χρειάζονται αυτά τα κονδύλια. Έστω και αν είναι περιορισμένα, καταλαβαίνετε και δεν αντικαθιστούν τις εθνικές παρεμβάσεις, συνδυάζονται ε, με, τις, ε, με εθνικές επιδοτήσεις. Η κυρία Λίν, ναι, δεν ήθελα να πάρω το λόγο, αλλά ακούγοντας τον κύριο Χέλμπερ δεν μπορούσα παρά να ζητήσω το λόγο. Ναι, δεν θα λύσουμε όλα τα προβλήματα, αλλά αφού το έχουμε το ταμείο, γιατί να μην το χρησιμοποιήσουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τώρα, να αλλάξουμε τους κανόνες ούτως ώστε κάποιοι που έχασαν τη δουλειά τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβουν κάποια βοήθεια έστω και μικρή για την επανακατάρτιση τους. Ε, έχουμε τα κονδύλια, πρέπει να μεριμνήσουμε τόσο ώστε να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για την εκ νέου κατάρτιση για όσους έχασαν τη δουλειά τους λόγω της οικονομικής ύφεσης. Όποια και αν είναι η απόψή σας, συγγνώμη, αλλά είναι σημαντικό να εγκριθεί σύντομα ε, ταχύτατα η τροποποίηση του κανονισμού για τους ε, ψηφοφόρους μας ε, που υποφέρουν γιατί έχουν χάσει τη δουλειά τους. Σας ευχαριστούμε. Δεν έχουμε κανέναν άλλον ε, που έχει ζητήσει το λόγο. Η Επιτροπή δεν θέλει, όχι, γνέφει αρνητικά. Η κυρία Στάουνερ, λοιπόν, ε, για να συνοψίσει τη συζήτηση η ενόψη της αυριανής ψηφοφορίας. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω εγκάρδια όλους τους συναδέλφους μου. Και μου φαινόταν στην αρχή εξαιρετικά περίπλοκος αυτός ο φάκελος. Τώρα όμως ε, έχουμε ένα ευτυχές τέλος, ελπίζω. Όπως σας είπα, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι μια σύντομη, γλίγορη διαδικασία, γι' αυτό απέστερα και όλες αυτές τις τροπολογίες. Ελπίζω ότι μπορείτε να συμφωνήσετε με αυτά τα τρία-τέσσερα σημεία που παρουσίασα προηγουμένως στην εισαγωγή μου, γιατί σας είπα και ξεκάθαρα ο στόχος είναι το ταμείο αυτό να είναι πιο αποτελεσματικό, πιο γλίγορο στις αντιδράσεις τους. Ο στόχος δεν ήταν να δημιουργηθούν κάποιες συμπληρωματικές δυσκολίες και έναντι της Κομισιόν. Δεν ήταν καθόλου αυτή η πρόθεσή μου. Το είδατε και στην αρχή της παρέμβασής μου, έτσι όμως νομίζω προχωρούμε πολύ καλά. Εξακολουθούμε να συνομιλούμε την Κομισιόν και το Συμβούλιο Ποια θα είναι τελικά η θέση τους δεν μπορούμε να το προβλέψουμε ακόμα. Αλλά νομίζω ότι η στάση μας είναι πάρα πολύ καλή. Προασπίζουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων και αυτός είναι ο στόχος μας νομίζω ως κοινωνική πολιτική στην Επιτροπή μας αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε άρα λίγη η συζήτηση. Θα ψηφίσουμε αύριο. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο σημείο. Ε, μέτρα για την ε, βελτίωση ασφάλειας κατά την εργασία των εγγύων λεχών και αλουφουσών εργαζομένων. Η επί της ουσίας αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή Γυναικών. Η δική μας εισηγήτρια της νομοδότησης είναι, η συντάκτη της είναι η κυρία Μαντέρα. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι μιλούσαμε για ενισχυμένη συνεργασία, αλλά ξέρετε ότι γνώρισε αυτή η έκθεση πολλές ε, περιπέτειες. Εντάξει. Ε, ε, ε, Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συνεισέφεραν σε αυτή τη συζήτηση και αυτή την έκθεση και ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες αυτές οι τροπολογίες και με βάση τη συζήτηση μαζί με την Επιτροπή ακολουθούμε παράλληλες πορείες και μπορούμε να πούμε ε, ότι συμβαδίζουμε ως προς το περιεχόμενο με την Επιτροπή σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα και σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν πάση περιπτώσει, κατά την εξέλιξη της κατάστασης προσπαθήσαμε να φτάσουμε σε συμβιβασμούς, αν και το θέμα δεν είναι και τόσο απλό γιατί η διάρθρωση της Επιτροπής είναι αρκετά απλή και οι επιλεκτικές, ε, οι εναλλακτικές λύσεις είναι πιο περίπλοκες. Εν πάση περιπτώσει είναι επικοδομητική η εργασία. Υπάρχουν ορισμένε ε, τροπολογίες που μπορούμε να πούμε ότι βρίσκονται κατά μέρος αυτής της ε, προοπτικής της Επιτροπής, ως προς την πλειοψηφία της και νομίζω ότι δεν έχουν άμεση σχέση με τις τροπολογίες Στάουνερ και Μαν. Αναφέρομαι στις τροπολογίες Τόμας Μαν, όπου θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες να τις εντάξουμε στο συνολικό πνεύμα της έκθεσης, διότι ότι βρίσκονται, δεν βρίσκονται μέσα στο πνεύμα που διέπει την Επιτροπή. Σε αυτή τη φάση θα ήθελα απλώς να πω σε σχέση με την τροπολογία 40, επειδή θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή διάρθρωση που να διέπει την πρόταση επιτροπή σε σχέση με την τροπολογία 40 θα ήθελα να ζητήσω από τη συνάδελφο Στάουνερ να την ε, καταστήσει πιο σαφή διότι είναι αξιέπαινη αυτή η στόχη αλλά δεν ξέρω κατά πόσο βελτιώνουν την πλαισίωση του θέματος. Θα ήθελα λοιπόν ορισμένες διασαφηνίσεις από τη συνάδελφο Στάουνερ για την ε, τροπολογία 40 για να δούμε πώς είναι δυνατόν μέχρι την αυριανή ψηφοφορία να επιλύσουμε το θέμα. Λαμβάνοντας υπόψη το πορτογαλικό κείμενο και κοιτώντας και το αγγλικό και γαλλικό κείμενο σε σχέση με τη δική μου τροπολογία 43 υπάρχει ένα λάθος σε σχέση με την προφορική ε, τροπολογία σε σχέση με μητέρες με αναπηρίες. Αυτό αφορά ένα συντακτικό θέμα του πορτογαλικού κειμένου. Νομίζω ότι τις περισσότερες γλώσσες ε, δεν θα έχει να τροπολογία έτσι όπως είναι διατύπωμένη. Το αγγλικό και γαλλικό κείμενο είναι σωστό. Και ίσως χρειάζεται μια προφορική τροπολογία για να διασαφηνίσουμε αυτό το κείμενο. Θα ήθελα η κυρία Στάουνερ να μας επεξηγήσει την τροπολογία υπαριθμών 40. Σας ευχαριστούμε κυρία Μαντέιρα. Μα ε, όντω υπάρχει ενισχυμένη συνεργασία για αυτή τη γνωμοδότηση. Κυρία Στάουνερ, μπορείτε να μας, Στάουνερ, μπορείτε να μας εξηγήσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι Μαδέρα, και η συγγετρία και εγώ Έχουμε τις ε, τροπολογίες 12 και 53 με τη βοήθεια των οποίων καταλήξαμε σε μια συμβαστική τροπολογία. Έχω υποβάλει και μια άλλη πρόταση για συμβαστική τροπολογία. Αυτή η κατανομή της ε, προστασίας μητέρα σε 2 εβδομάδες πριν από, την, ε, από το τοκετό και η ψή μετά το δοκιτό είναι μια ε, συμβαστική πρόταση της 37 Μαδέρη και 40 της δικής μου νομίζω ότι θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε πως αυτά γιατί θεωρούμε και οι δύο ότι εάν όπως θέλει η Κομισιόν αφήνουμε τελείως ανοιχτή αυτή την κατανομή της περίοδου προστασίας της μητέρας πριν και μετά το, το, και οι εργοδότες καμιά φορά ασκούν πίεση στην έγκυο γυναίκα εργαζόμενη να πάρει όλη την άδεια μετά, μετά το τοκετό. Πράγμα που ε, καμιά φορά όμως είναι λογικό να έχει και μερικές εβδομάδες πριν από το τοκετό η γυναίκα αυτή την ελόγω προστασία. Και γι' αυτό θεωρώ ότι μπορώ να συμφωνήσω καταρχήν με την ε, τροπολογία 37 της εισηγητρίας. Έχω υποβάλει μια σχετική τροπολογία συμβαστική δική μου, αλλά δεν έχω ακούσει την αντίδραση της εισηγητρίας. Θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε το θέμα. Και μετά πρέπει να δούμε τη δική μου τροπολογία 48. Αγαπητοί συνάδελφοι, μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι προθεσμίες προστασίας απόλυσης να μην τελειώνουν όταν τελειώσει η περίοδος προστασίας, αλλά λίγο παραπάνω. Γιατί κάθε εργαζόμενη γυναίκα, και εγώ είμαι μια εργαζόμενη γυναίκα, όταν επιστρέψει κανένα στην εργασία του μετά από την περίοδο προστασίας, τις πρώτες εβδομάδες έχει κάποια προβλήματα με το τι θα γίνει με το παιδί, θα πρέπει να φύγει πιο νωρί από τη δουλειά για να πάει να το πάρει το παιδί από το προβοληπιακό σταθμό. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει καμία προστασία, ακριβώς ο εργοδότης τις δύο ε, ή παραπάνω πρώτες εβδομάδες μέχρι να λυθούν αυτά τα αρχικά προβλήματα ίσως απολύσει. Γιατί εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει η προστασία από απόλυση να είναι τέσσερις μήνες μακρύτερη από την ε, περίοδο προστασίας. Και γι' αυτό το έχω πει και το ξαναλέω. Το ότι έχει προσθεθεί το όνομά μου στις τροπολογίες του συναδέλφου Μαν δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Είναι ένα πρόβλημα της ε, γραμματείας. Εκτός από την κοινή τροπολογία 55, εγώ δεν συμμερίζομαι καμία από τις τροπολογίες του συναδέλφου Μάν. Σας το λέω ξεκάθαρα. Δυστυχώ έγινε κάποιο σφάλμα, αλλά δεν φταίω εγώ. Και δεν μπορούσε φαίνεται να αλλάξει κιόλα. Λοιπόν, υποστηρίζω και αυτή είναι και η μορφή της δικής μου στην ομάδα εκτός από την τροπολογία 55 καμία από τις τροπολογίες Τόμας Μαν. Αυτό το ξέρει και η συγκέντρια νομίζω. Γιατί αυτό θα ήταν αντίθετο με τη γραμμή που ακολουθώ γενικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριος Μπούσελ Μάθιος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να πω κάτι για την ε, συμβαστική τροπολογία Β που λέει ότι τα κράτη-μέλη θα μεριμνήσουν ούτω ώστε η χρήση τη άδεια της μητρότητας ε, δεν θα πλήξει την ε, επιχειρήση κτλ. Δύο παρατηρήσεις γι' αυτό. Πρώτον, ποιο είναι ο στόχο αυτή τη συμβαστική τροπολογία μέσα σε αυτή τη γνωμοδότηση. Αν δεν κάνω λάθο, ε, η γνωμοδότηση είναι περί τη βελτίωση τη ασφάλεια και τη υγεία στον χώρο τη εργασία για τι εγγύου, για τι λεχόνε και για τι θυλάζουσε. Δεν έχει καμία σχέση με την υγεία και την ασφάλεια αυτή η τροπολογία. Δηλαδή πρόκειται για την πνευματική ηρεμία των ανθρώπων, ναι μεν, αλλά δεν είναι το αντικείμενο τη νομοδότησή μα. Αλλά προτιμώ να καταργηθεί αυτή η συμβιβαστική τροπολογία γιατί δεν είναι η θέση τη μέσα στην νομοδότηση. Όμω, αν η, ε, κρίνει η συγγήτρια, και εφόσον αυτή είναι η συγγήτρια, κρίνει ότι πρέπει να τη συμπεριλάβουμε, τότε θα ήθελα να προτείνω να αλλάξουμε την διατύπωση έλαφρω με μια προφορική τροπολογία, διότι αν δεν κάνω λάθος, το κοινοβούλιο δεν μπορεί να επιβάλλει τι πρέπει να κάνουν και δεν πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη για τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Τα κράτη-μέλη μπορούμε να πούμε θα μεριμνήσουν ούτω ώστε να και τα λοιπά. Γιατί πρόκειται για εθνική αρμοδιότητα όταν μιλάμε για τα ε, συντάξιμα ε, ε, δικαιώματα για συνταξιοδότηση. Οπότε προτείνω στην εισηγήτρια και στους συναδέλφους μια προφορική τροπολογία που θα λέει θεωρεί ότι τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να εξασφαλίσουν ότι η χρήση της άδειας μητρότητας δεν επηρεάζει τα συντάξιμα δικαιώματα. Ε, νομίζω ότι είναι πιο σωστό. Σας ευχαριστώ. Η εισηγήτρια θέλει το λόγο για να σχολιάσει παρεμβάσει των συναδέλφων. Ευχαριστώ σε σχέση με τα θέματα που έθιξε η κυρία Σάουνερ στη τροπολογία 48 μετά από την άρση των αμφιβολιών θεωρώ ότι μπορεί να γίνει αποδεκτή και μπορούμε να τη δεχτούμε. Σε σχέση τώρα με την τροπολογία 40 θεωρώ ότι θα πρέπει μέχρι την τροπολογία, να, μέχρι την ψηφοφορία με συγχωρείτε, να το δούμε το ζήτημα αλλά θα πρέπει να δούμε κατά πόσο ορίζουμε κατόφλια ή ανώτατα όρια. Ε, γιατί εδώ υπάρχουν και ζητήματα αρχής και βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος, μπορώ να πω με την Επιτροπή. Και εδώ μιλάμε για λεπτομέρειες κυρίως. Σε σχέση με τα δικαιώματα συνταξιοδότησης είναι σαφές ότι τα δικαιώματα αυτά δεν αποτελούν θέμα. Η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία σχετικά σχετίζεται με την προστασία που παρέχει το κράτος προνοίας. Εμείς δεν αναφερόμαστε στα διάφορα συστήματα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα θέμα αρμοδιότητας, κρατικής αρμοδιότητας, αλλά πρόκειται για ένα ελάχιστο δεν τα αφήγουμε όποιο και να είναι το σύστημα που ισχύει στα κράτη-μέλη. Αυτό είναι θέμα κοινοτικού συμφέροντος, συμφέροντος του εργαζομένου για την ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας του, διότι σε σχέση με τις ώρες και τύπο εργασίας έχει μεγάλη σημασία. Άρα δεν είναι παράπλευρο το ζήτημα. Γνωρίζουμε ότι σήμερα έχει μεγάλη σημασία για το μέλλον μας για να έχουμε δίκτες ε, φτώχειας όταν μιλάμε για γυναίκες και για ηλικιωμένους. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή πλαισίωση ως προς τον δημόσιο τομέα και δεν θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν αυτές, αυτή η κατάσταση για το μέλλον. Αυτό είναι ύψης της σημασίας και θα πρέπει να το καταστήσουμε σαφές για να προσαρμοστούν και τα διάφορα εθνικά συστήματα. Αυτή είναι μια σύσταση, τίποτα παραπάνω. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι μια σύσταση με βάση ένα κατόφλι που ορίζουμε και όχι ένα ανώτατο όριο. Δεν ξέρω κατά υπάρχει διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης. Ευχαριστώ. Κύριε Σουσάτερ, ζητήσατε το λόγο. Έχω τελειώσει τη συζήτηση. Θα σας δώσω το λόγο, αλλά είχα δυνατότητα να πάρετε το λόγο προηγουμένως, πριν να το δώσω στην εισηγήτρια. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Μία ερώτηση ήθελα να υποβάλω. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς γιατί απορρίπτει την τροπολογία 21. Μήπως μπορεί να μας το εξηγήσει η συγχύτρια. Ωραία. Άρα θα ξαναδώσουμε το λόγο στην κυρία Τζαμέλα. 31. Τροπολογία 21. Σε σχέση με την 21, δεν ξέρω κατά πόσο ο κύριος Μπούσιλ Μάθιος ήδη έθιξε το ζήτημα. Ε, είπα ότι δεν μιλάμε εδώ για δικαιώματα συνταξιοδότησης. Σε αυτή την περίπτωση ίσως αντιμετωπίσουμε θέματα ένταξης. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να ενσωματωθούν εδώ, να περιληφθούν εδώ. Αλλά και η 58 αναφέρεται στο ίδιο και την έχουμε εντάξει. Και επιτρέπει την χρήση με την ίδια λογική που διέπει την 21. Δηλαδή μπορούν οι ενώσεις, οργανώσεις και ε, λοιποί νόμιμοι φόρεις να ε, διέπουν την ίδια, να διέπονται από την ίδια πλαισίωση είτε πρόκειται για την 21 είτε για την 58. Η 58 όμως έχει συνταχθεί καλύτερα και νομίζω ότι προστατεύει τις γυναίκες ε, καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ. Άρα λίγη και η συζήτηση του θέματος αυτού. Θα γίνει η ψηφοφορία αύριο όπως γνωρίζετε και τώρα θα ασχοληθούμε με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας. Jean Lambert. Uh, um, Ευχαριστώ, Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους διάφορους συναδέλφους που υπέβαλαν τροπολογίες. This report, um, not least for the content of many of those... Και ιδίω όσον αφορά το περιεχόμενο των τροπολογιών αυτών. Καθώ επίση και για τη συνεργασία που είχαν στη... σχετικά με το κατάλογο τη πληροφορία για να βρεθούν κάποιοι συμβιβασμοί. Καταφέραμε να βρούμε μια σειρά συμβιβασμών την Α παραδείγματο χάρη στην βασική τροπολογία που αφορά του κοινωνικούς ε, βοηθούς και τις δραστηριότητες στην αγορά εργασίας στη βασική τροπολογία Β για τις κοινωνικές υπηρεσίες και γενικά υπηρεσίες γενικού συμφέροντος ε, τροπολογία Δ όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση ε όσον αφορά τον οδικό χάρτη για την ενεργό συμπερίληψη που προβλέπει τώρα πια την ένταξη των τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε κάποιες άλλες επίσης όπως η ΓΑΜΑ που αφορά την νομοθεσία κατά των διακρίσεων. Μπερέσαμε να βρούμε και ένα συμβασμό για τη ΓΑΜΑ όσον αφορά την εφαρμογή του σών διατάξεων για την υπάρχουν διαφορετικέ ε, απόψει για το τι θα κάνουμε για διαφορά. Με συγχωρείτε, πώ μπορείτε να σταματήσετε να μιλάτε εδώ δίπλα μου. Βέβαια, αυτό σχετίζεται και με αυτό που ψήφιζαμε την ε, Πέμπτη. Η γραμμή που ακολούθησα σε διάφορου συμβασμού είναι εκεί που ειδικά ε, ορισμένα τμήματα μια, τμήματα θα περάσουν σαν προφορικέ τροπολογίε. και πρότεινα να κάνουμε κάτι που να μην έχουμε μια προφορική τροπολογία που μπορεί να είναι θύμα ενός βουλευτή. Όσον αφορά λοιπόν την ε, επέκταση της νομοθεσίας έχουμε την ε, τροπολογία 79 ΛΙΝ που είναι υπέρ αυτής της ε, διεύρυνσης. και νομίζω ότι είναι καλύτερη από το τρίτο τμήμα της τροπολογίας 88 που θα ήταν τελικά προφορική προσθήκη. Καμιά φορά ίσως ε, έχουμε την εντύπωση ότι το αποτέλεσμα θα ήταν κάπως ατυχές στην εντύπωσή του γιατί θα, ήταν ορισμένες, θα είχε ορισμένες επικαλύψεις κλπ. Αλλά νομίζω ότι φέρνουν καλύτερα παρά από το να περάσουμε από προφορικές τροπολογίε που δεν μα αρέσουν και πάρα πολύ. και μπορέσαμε νομίζω να συμφωνήσουμε και να συμβαστούμε όσον αφορά τις ευάλωτες ομάδες. Διαγράψαμε με τον ορισμό που υπήρχε στις αιτιολογικές σκέψεις για να εξετάσουμε πολύ καλά από την τροπολογία 66. Ε, μετά προσπαθήσαμε να έχουμε μια συμβιβαστική πρόταση γύρω από την τροπολογία 6 για την προτινόμενη οδηγία. Δεν έχουμε όμως κανένα συμβιβασμό. Δεν απορρίεται σίγουρα. Αυτό που έχουμε τώρα είναι μια επιλογή ναι ή όχι όσον αφορά την παράγραφο αυτή στο κατάλογο ψηφορίας και ο όποιος θέλει να το διαγράψετε. Υπάρχουν άλλε επιλογέ για την αντικατάστασή του. Σε σχέση και με το Ευρωπαϊκό Έτο κατά τη φτώχεια. Ένα από τα άλλα θέματα Income. Um, Μετά θα ήθελα να δούμε τα, τις τροπολογίες που αφορούν την επαρκή υποστήριξη του εισοδήματος, όπως το αναφέρει και η σύσταση της Κομισιόν και του Συμβουλίου. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να ανεκαταστήσει κανείς κάποια τμήματα του κειμένου εδώ. Γιατί κάποιε από τροπολογίε που δίνουν την εντύπωση ότι είναι ευθυγραμμισμένε συμπεριλαμβάνουν και άλλε ιδέε που σημαίνουν ότι δεν αλλάζουμε πραγματικά μία διατύπωση και θα ανακαστούμε από μία άλλη διατύπωση. Έχουμε ας πούμε την παράγραφο 5, παράγραφο 6 κλπ. Αλλάζουμε όμως με τροπολογίες τελείως την φύση των παραγράφων αυτών. Η τροπολογία 34 της ε, Άνφαν Λάγκερ ήταν χρήσιμη γιατί ορίζει τι εννοούμε όταν λέμε επαρκές επίπεδο εισοδήματος. Αυτά με δύο λόγια όσον αφορά τις συμβαστικές προτάσεις. Είπαμε η υποστήριξη του εισοδήματο και όχι ελάχιστο εισόδημα, αλλά όπω σα είπα είναι πολύ εξυπηρετική εδώ η τροπολογία 34 τη Αλβαν Λάγκερ. Και αυτά είναι τα σημεία στα οποία θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή των συναδέλφων και να επαναλάβω τι ευχαριστίε μου για τη συνεργασία. Παρόλο που σα δεν πετύχουμε συνένεση, η συνεργασία ήταν πάρα πολύ θετική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πριν ναι, ακούσουμε τους ομιλητές, έχουμε το κύριο... Έχουμε 9 εκπροσώπους από το Εθνι... Συνδικάτο, Ευρωπαϊκό Συνδικάτο και από το Αλληλεγγύης. Η κυρία Λίν και ο κύριος ε, Μπούσελ Μάθιος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Τζιν για τη συνεργασία. Ευχαριστώ που ανέφερες ότι θα υποστηρίξεις τις τροπολογίες μου για την υποχρεωτική ηλικία συνταξιοδότησης και τα λοιπά όλες τις τροπολογίες που υπέβαλα. Η μόνη διάσταση απόψεων νομίζω που υπολείπεται είναι σχετίζεται με το ελάχιστο εισόδημα. Είμαι υπέρ του ελάχιστου εισοδήματο που θα προσδιορίζεται σε εθνικό επίπεδο, το γνωρίζει Αυτό είναι σημαντικό να προσδιορίζεται από τα κράτη-μέλη. Απλά με δυσκολεύει το εξή και το γνωρίζω ότι όταν προτείνει μια συμβαστική τροπολογία ουσιαστικά μιλά για ελάχιστο εισόδημα και μια οδηγία για το ελάχιστο εισόδημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν νομίζω ότι είναι ε, η σωστή κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε. Προσπαθήσουμε να πείσουμε όλα τα κράτη-μέλη δηλαδή να αναπτύξουν δικό του σύστημα ελαχίστου εισοδήματος. Ε, τώρα για την τροπολογία 34 της ε, Anfan Lanker. Καλή είναι η πρόταση και πρέπει να την υποστηρίξουμε κατά τη γνώμη μου γιατί δεν λέει ότι πρέπει να το προσδιορίσουμε σε κοινοτικό επίπεδο, λέει ότι καταρχάς είμαστε υπέρ του ελάχιστου εισοδήματο για να ε, εξασφαλίσουμε ότι δεν θα ζουν κάτω από το όριο της ε, φτώχειας ε, οι πολίτες, δηλαδή θα έχουν τα ζήν, θα ξεφύγουν από τη φτώχεια και κατά τη γνώμη μου όλοι σε αυτό αποσκοπούμε. Μπορώ να την υποστηρίξω αυτή την ε, τροπολογία λοιπόν και ε, νομίζω και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Χωρίς να επιδιώκουμε οπωσδήποτε να γίνει κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι σημαντικό να έχουμε την ευρύτερη δυνατή συνένεση για αυτό το θέμα, όπως ακριβώς και για τα θέματα της κατάργησης, της διακριτικής μεταχείρισης που έχω βάλει στις τροπολογίες μου. Αποκλείονται διάφοροι από διάφορες ε, διάφορους τομείς της ζωής, ε, διότι έχουν αναπηρίες ή έχουν άλλη ηλικία, έχουν άλλες, ε, άλλο σεξουαλικό προσανατολισμό, άλλες θρησκευτικές πεπιθήσεις και σε όλες τις νομοδοτήσει εγώ ε, που σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη και τον κοινωνικό αποκλεισμό, το προτείνω αυτό στις τροπολογίες μου, θέλω να εξασφαλίσω ισότιμη μεταχείριση, δεν θέλω να αποκλείεται κανένας και να μην έχει ένα αποδεκτό πρότυπο διαβίωσης, αλλά όχι μόνο και πρόσβαση σε, ό,τι δικαιούται και ευχαριστώ πάρα πολύ που με υποστηρίζεις ε, για αυτή την τροπολογία. Ξέρω όμως ότι υπάρχει διάσταση απόψεων για αυτό το θέμα, όχι μόνο στην Επιτροπή μας, αλλά και γενικότερα στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Μπούσελ Μάθιος και η κυρία Παναγιωτοπούλου Κασιώτο ακολουθούν. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Ε, η πολιτική μου ομάδα είναι υπέρ της ενθάρρυνσης, της παρακίνησης προς τα κράτη-μέλη να ορίσουν ένα ελάχιστο εισόδημα, αλλά κατά τη οδηγίας. Δεν πρόκειται ποτέ να περάσει μια τέτοια πρόταση από το Συμβούλιο, οπότε δεν αξίζει να ακολουθήσουμε αυτή τη ρότα. Απλά να το τονίσουμε αυτό το βασικό μήνυμα. Ε, Τζιν, ξέρω ότι δεν σα αρέσουν οι προφορικέ τροπολογίε. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα υποβάλω μια προφορική τροπολογία. Σε παρακαλώ να την εξετάσει. Στην τροπολογία Β, στη, στη μέση περίπου, που λέει για το, την Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο. Η πρόταση που λέει knows that progress must be made και τα λοιπά για τις καθολικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες κοινής ωφελίας δεν με προβληματίζει η ίδια η πρόταση, απλά με προβληματίζει αρκετά ώστε να κάνω μια πρόταση. Γιατί λέμε στην αρχή τη πρόταση. Ε, σημειώνει ότι πρέπει να σημειωθεί πρόοδο, λέει τώρα το κείμενο. Μα γενικότερα αυτό είναι γεγονό. Ναι, όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να σημειωθεί πρόοδο. Δεν. Ε, Συμφωνούμε όμως απαραίτητα για το γεγονός ότι η απάντηση είναι να αναπτύξουμε ένα σχέδιο δράσης σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Μπορεί να φτάσουμε σε αυτό, να θεωρήσουν όλοι ότι αυτή είναι η απάντηση, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι σημειώνει ότι αυτή είναι η απάντηση. Επ' αυτού δεν υπάρχει συμφωνία, οπότε προτείνω το πρώτο κομμάτι της πρότασης να μείνει ως έχει, ότι ε, σημειώνει ότι πρέπει να σημειωθεί πρόοδος και μετά να αναφερόμαστε στις υπηρεσίες κοινή ωφελίας να πούμε και θεωρεί ότι η ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης ε, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Οδηγίας πλαίσιο για την κατοχήρωση αυτό είναι η, ε, ε, η βέλτιστη προσέγγιση. Για να μην υπάρχει αυτή η παρανόηση που σας εξήγησα. Ε, Επίση ε, μιλάμε για κατοχήρωση των υποχρεώσεων για τι καθολικέ υπηρεσίε. και στο δεύτερο κομμάτι λέμε για κατοχήρωση δικαιωμάτων αλλά άλλο υποχρέωση παροχής υπηρεσία, υπηρεσίες ε, γιατί αυτό αφορά τον πάροχο και άλλο υποχρέωση το δικαίωμα μάλλον του δικαιούχου. Πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό αφήνοντα όμω αναλύωτο το βασικό μήνυμα. Ελπίζω αυτή τη φορά να κάνει μια εξαίρεση τζιν και να τη δεχτεί την προφορική τροπολογία που υποβάλλω. Ευχαριστώ. Η κυρία Πανάγιοτοπούλου Κασιώδη και η κυρία Φανλάκεν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και βέβαια ε, συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι για ένα τόσο σπουδαίο θέμα που είναι η ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα ε, στην αγορά εργασίας πρέπει να, έχουμε, να βρούμε ε, κοινή γραμμή και με την ευκαιρία και του έτους κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού να δώσουμε ένα μήνυμα ε, προς ε, τους Ευρωπαίους πολίτες ότι σε αυτό το θέμα ε, θα έχουμε όλοι μαζί σύμπνοια και κοινούς στόχους. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα καλό κείμενο, χωρίς περιττές επαναλήψεις. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάθε φορά να αναφέρουμε ε, το ε, ότι έχει αποφασιστεί με οδηγίες. Ε, την μη διάκριση την έχουμε αρκετά τονίσει σε προηγούμενες οδηγίες. Γιατί πρέπει κάθε φορά να την επαναλαμβάνουμε. Γιατί πρέπει να επαναλαμβάνουμε την καταπολέμηση της βίας, της οικογενειακής βίας ή τα ναρκωτικά ή άλλα θέματα που χάνουν τον κοινό στόχο ε, και ε, γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει ε, με την ψηφοφορία μας να καθαρίσουμε λίγο το κείμενο. Επίσης για το ελάχιστο εισόδημα και στην έκθεση του Κοινοβουλίου για το έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού είχαμε αρκετά τονίσει ότι δεν είναι μόνο το εισόδημα εκείνο που έχει σημασία. Έχει σημασία η συνολική δυνατότητα να ζήσει κανείς μέσα σε αξιοπρεπείς συνθήκες και το εισόδημα είναι ε, ένας από τους παράγοντες. Αν όμως λείπουν άλλοι παράγοντες τότε ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε επιτελέσει το στόχο μας. Ε, γι' αυτό και μιλούμε για επαρκή εισοδηματική υποστήριξη, όπως μιλάει και το Συμβούλιο και νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε αυτή την κοινή γλώσσα, να μιλούμε για το θέμα αυτό με έναν μόνο όρο έχοντας ένα κοινό στόχο που δεν είναι διαφορετικός και που πρέπει να ε, είναι ε, υπεύθυνο το κράτος μέλος να τηρήσει αυτό το στόχο της επαρκούς εισοδηματικής υποστήριξης ε, ανάλογα με τα δικά του δεδομένα ε, και όχι βάσει οδηγίας όπως τονίστηκε και από τον κύριο Μπούσιλ Μάθιος, ε, Αν επιμείνουμε σε ιδεολειψίες θα χάσουμε τον κύριο στόχο μας που είναι η ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας. Ε, ελπίζω λοιπόν ότι ε, θα ε, καθαρίσουμε την οδηγία από περιτά και υποστηρίζοντας και τις συμβιβαστικές τροπολογίες εκτός από εκείνη που αναφέρεται στην εκπαίδευση μια και η εκπαίδευση είναι ένα θέμα αρμοδιότητας των κρατών μελών θα έχουμε τελική σύμπνοια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Η, κυρία Φανλάκη και η κυρία Τσίμερ ακολουθούν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ε, ήθελα να ζητήσω από την Τζίν να μου πει ε, ποια είναι η προσέγγιση που ακολουθεί για το ελάχιστο εισόδημα. Αλλά ρυθμίστηκε μάλλον το θέμα γιατί με την τροπολογία 34 αναφερόμαστε ήδη στο ελάχιστο εισόδημα. Φιστώ την προσοχή των συναδάλφων στο ότι πρόκειται για εθνική αρμοδιότητα. Το κράτος μέλος θα ορίσει ποιο είναι το ελάχιστο εισόδημα, οπότε δεν συνεπάγεται ότι θα υπάρξει σε κοινοτικό επίπεδο προσδιορισμός του ελαχίστου εισοδήματος. Είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μου επιτέλους να ε, ολοκληρώσουμε αυτήν την ε, ατελείωτη συζήτηση για το ελάχιστο εισόδημα και η κυρία Πούλου Κασιώτου έχει απόλυτα δίκιο όταν σχολιάζει αυτό το θέμα. Η κυρία Λίν διορθώνει την αγγλική διερμηνία, μιλάμε για ελάχιστο εισόδημα και όχι για ελάχιστο μισθό, έτσι. Ε, για ελάχιστο εισόδημα μιλούσα εγώ, ούτως ή άλλως δεν μιλούσα για ελάχιστο μισθό. σε κάποια κράτη-μέλη μπορεί να πρόκειται όντω για ελάχιστο μισθό. Αυτό είναι ένα γεγονός στο Συμβούλιο Υπουργών δεν καταφέραν ποτέ να συμφωνήσουν για ένα ευρωπαϊκό ελάχιστο εισόδημα. Μπορεί να υπάρξει κάποιος ρόλος για την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσδιορίσει ποια είναι τα εισοδήματα που επιτρέπουν μια αξιοπρεπή διαβίωση ε, για τους πολίτες. Και συμφωνώ με την ε, κυρία Παναγιωτοπολου Κασιώτου που μας λέει ότι δεν είναι θέμα εισοδήματος μόνο η φτώχεια. Υπάρχει η πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες. Υπάρχουν και άλλες διαστάσεις πολύ σημαντικές για όσους ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Είμαι πεπισμένη όμως ότι αν δεν ε, ε, υπάρχει ένας μισθός ε, που είναι, αντιστοιχεί το 50% του μεσαίου εισοδήματος της χώρας στην οποία διαμένει το εν λόγω άτομο, δεν μπορεί να ξεφύγει κάποιος από το, τη φτώχεια. Ευχαριστώ την Τζιν Λάμπερτ. Ήταν εξαιρετική η συνεργασία που είχαμε και καταλήξαμε τελικά σε αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες και περιμένουμε την αυριανή ψηφοφορία. Η κυρία Τσίμερα, αλλά πρώτα θέλω να πω... Και στα Σουηδικά υπάρχει ένα προβληματάκι με αυτή την ορολογία, ελάχιστος μισθός, ελάχιστο εισόδημα. Στα Σουηδικά ε, ο μισθός προσδιορίζεται από τους κοινωνικούς εταίρους. Το ελάχιστο εισόδημα είναι το αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης βάσει των συστημάτων ε, κοινωνικής ασφάλισης. Σε τοπικό επίπεδο προσδιορίζεται αυτό στη Σουηδία και υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο μισθό και στο εισόδημα. Κυρία Λίν, Σίγουρα, είμαι σίγουρη ότι η κυρία Άνφαν Λάγκεν μιλούσε για ελάχιστο εισόδημα και όχι για ελάχιστο μισθό, ότι τους διερμηνείς διόρθωνα, γιατί ήθελα να το διευκρινίσω για να του ενημερώσω ότι μιλάμε για ελάχιστο εισόδημα και όχι για ελάχιστο μισθό. Κυρία Τσίμερ. Λοιπόν, το θέμα του ελάχιστου μισθού και του ελάχιστου εισοδήματο είναι κάτι που μας απασχολεί εδώ και πολύ καιρό και με ε, εκθέσεις που είχαμε τους περασμένους μήνες στην ε, Επιτροπή μας εδώ. Σας υπενθυμίζω τη συζήτηση που είχαμε στην αρχή της συζήτησης για την έκθεση Τζιν Λέμπερ όταν ένας από τους συναδέλφους είπε ότι όλο τα ίδια θέματα συζητάμε και δεν προχωράμε καθόλου. Και αναρωτήθηκε ποιο είναι το νόημα αυτής της ε, δράσεις. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω η Τζιν Λάμπερ για την εργασία που έχει επιτελέσει που μπορέσαμε και εδώ στην Επιτροπή μα να επαναλάβουμε τις θέσεις μας πολλές φορές για κάποια συγκεκριμένα θέματα. Ε, καμιά φορά δεν χρειάζεται, τα έχουμε πει πολλές φορές, αλλά ακριβώς αυτά τα πράγματα τα οποία δεν είναι η συνήθις πρακτική στην ευρωπαϊκή πολιτική και που θεωρούνται η βάση και στην Κομισιόν και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χρειάζεται, λέω, να τα ορίσουμε. Και γι' αυτό υπέλαβα εγώ κάποιες τροπολογίες που αναφέρουν σε θέσεις που έχουμε πάνω σε μια έκθεση της Επιτροπής αυτής με μια πλειοψηφία δύο τρίτων στην Ολομένη. Και ξέρουμε ότι όσον αφορά την μεγάλη σύγχυση που υπάρχει με το ελάχιστο εισόδημα, τα ελάχιστα συστήματα ασφάλισης και τους ελάχιστους μισθούς πρέπει συνεχώς να εξηγούμε και να ξαναεξηγούμε τι εννοούμε. Και θα ήθελα για άλλη φορά να τονίσω ότι γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικές τροπολογίες. Να πούμε ναι, ελάχιστη μεστή, ελάχιστα συστήματα ασφάλισης είναι εθνικό θέμα και υπάρχουν διαφορές στο πώς ορίζονται και πώς καθορίζονται στα κράτη-μέλη. Απ' την άλλη μεριά όμως θα πρέπει να είναι σαφές ότι κάθε ελάχιστος μισθός ή κάθε ελάχιστο σύστημα ασφάλισης που υπάρχει σε ένα κράτος μέλος αποτρέπει τους πολίτες να πέσουν στην φτώχεια. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει και ένα στοιχείο ποιότητας που ε, θα λέει ότι αυτή η μισθοί και τα συστήματα ασφάλισης δεν θα πρέπει να οδηγούν στη φτώχεια αυτή και αυτό πρέπει να το κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λέμε ότι θα χρειαζόμαστε αυτά τα πρότυπα. Θα πρέπει να υπάρχουν πρότυπα για την αντίσταση στη φτώχεια. Και έχουμε ορίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση από πότε υπάρχει ο κίνδυνος οι πολίτες να περάσουν στη φτώχεια για το ελάχιστο εισόδημα είναι στο 60% του εθνικού εισοδήματο του νοικοκυριού. Και όσον αφορά του μισθού, είναι στο 60% του μέσου όρου του εθνικού εισοδήματο, του εθνικού μισθού, συγγνώμη. Πάντα λοιπόν πρόκειται για θέματα <clears throat> εθνικά. Αυτό θα πρέπει να το ξέρουμε και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε για άλλη μια φορά και μέσα στα πλαίσια αυτής της έκθεσης. γιατί δηλαδή, έτσι μπορούμε να υποστηρίξουμε την Κομισιόν με τη σκέψη σας το τι πρέπει να κάνει, τι μπορεί να κάνει, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ορίσουμε κοινού στόχους για τα καταπολέμηση της φτώχειας και να μπορέσουμε οι μέθοδοι συντονισμού να ε, γίνουν αύριο πολιτικές. Και αυτό σας παρακαλώ να υποστηρίξετε τις τροπολογίες που είχα υποβάλει, ιδίω στις 42, 46, 47, 62, 80, 113, Πρόκειται για διατυπώσεις που είχαμε κάποια στιγμή αποφασίσει εδώ στην Επιτροπή και που είχαν περάσει με πλειοψηφία δύο τρίτων στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Τομασεύσκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να θίξω το θέμα που μόλις έδειξε και η κυρία Τσίμερ δηλαδή ένα κίνητρο για την ρύθμιση του, ελάχιστο, του ελάχιστου εισόδηματος στα κράτη-μέλη. Αλλά στις περισσότερες χώρες υπάρχουν αυτοί οι κανονισμοί σε σχέση με το ελάχιστο εισόδημα, διότι είναι κάτι που ρυθμίζει το κράτος. Καθώς και άλλες πτυχές της νομοθεσίας, το ζήτημα είναι πόσο λαμβάνει κάθε μέλος της οικογένειας. Αυτό είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό και γι' αυτό μιλάμε για αξιοπρεπή ποιότητα ζωής σε κάθε οικογένεια. Νομίζω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε μια οδηγία πλαίσιο όπως ορίζει και η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Χάρτα. Και μιλάμε για κατακεφαλή εισόδημα, όπου γίνεται λόγος για κατακεφαλή εισόδημα ή μέσο εισόδημα σε κάθε χώρα. Αυτό θα ήταν το καλύτερο δυνατό σε σχέση με αυτά που είπε και η κυρία Τσίμερ καθώς και η τροπολογία 46 σε σχέση με την ενεργό συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Είναι πολύ δύσκολο να πει κανεί ότι έχει καλή ε, ποιότητα ζωής εάν δεν μπορεί κανείς να ζει καλά από αυτά που κερδίζει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Δεν υπάρχει άλλος ομιλητής, οπότε η κυρία Λάμπερτ, παρακαλώ συνοψίστε. Σας ευχαριστώ. Um, Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους ε, συνεισέφεραν στη συζήτηση. Πολύ χρήσιμα θέματα εφήγησαν. Σε σχέση με την τροπολογία Β, δεν είναι δική μου η απόφαση, αλλά είναι και απόφαση άλλων, οι τροπολογίες των οποίων ε, ενσωματώνονται επίσης. Γι' αυτό νομίζω ότι και η προφορική τροπολογία του Φίλιπ δεν ρυθμίζει το πρώτο τμήμα αυτής της τροπολογίας συμβιβασμού, αλλά μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά. Τώρα, σε σχέση με το ρόλο των κρατών μελών, έναντι της Επιτροπής, Νομίζω ότι καθίσταται σαφές ότι τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για, τα, για την θέσπιση ορίων και την καταβολή των, του εισοδήματος, αλλά και στη ρύθμιση του Συμβουλίου που είναι η πιο ήπια νομοθεσία, η Επιτροπή συμπεριλαμβάνει αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές. Άρα δεν πρόκειται για απόλυτο διαχωρισμό αν και η έμφαση δίδεται στα κράτη-μέλη. Και καταλαβαίνω ποια θα είναι η τύχη της παραγράφου 6 ως προς την οδηγία πλαίσιο, αλλά μπας περιπτώσει το προσπαθούμε έτσι κι αλλιώς. Προβάλλουμε ιδέες και θα δούμε κατά πόσο θα επιθυστούν ή θα επιπλέψουν. Έχει υπάρξει μια συμφωνία σε σχέση με τα όρια ε, διαβίωσης, τέτοιας διαβίωσης έτσι ώστε να μην βρίσκεται κανείς στο κατόφλι της φτώχειας. Και ως προς την κατάρτιση, αυτό που έχει σημασία είναι η χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και άλλων μέσων για να ορίσουμε ε, την κατεύθυνση τη γενική κατεύθυνση, άρα δεν μπορούμε παρά να συμμετέχουμε ενεργά σε αυτόν τον καθορισμό των προτεραιοτήτων για τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Άρα βλέπουμε που προς τα που η πλειοψηφία. Θα κάνω κάτι για τροπολογία Β, αλλά δεν υπόσχομαι τίποτα γιατί δεν θα συμφωνήσω, δεν πρόκειται για δική μου απόφαση αποκλειστικά. Σας ευχαριστούμε. Αύριο θα ψηφίσουμε και για αυτή την γνωμοδότηση. Λίγη συζήτηση τώρα. Σημεία 8 και 9 τώρα. Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και το σχετικό προαιρετικό πρωτόκολλο που επισυνάπτεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Η κυρία Γέλεβα είναι η συγγήτριά μας και της δίνουμε αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους συναδέλφους που υπέβαλαν ε, τροπολογίες και να ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερως ε, τους σκιώδεις εισηγητές και θα ήθελα να τονίσω ότι πρόκειται ε, για την πρώτη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών στην οποία θα ε, προσχωρήσει επίσημα η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα γίνει συμβαλόμενο μέρος για αυτό το θέμα, για τα άτομα με αναπήρεια. Σας ε, διαβεβαιώ ότι για μένα δεν πρόκειται απλά για ε, ένα, μια δουλειά που κάνω, μια γνωμοδότηση που συντάσω. Είμαι πεπισμένη ότι πρέπει να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματα ε, των ατόμων με αναπηρία. Υπάρχουν ε, ήδη πολλές χώρες που έχουν γίνει συμβαλόμενα μέρη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Σουηδία, η Γερμανία, ε, σχάτως η Ιταλία, στις 3 Μαρτίου η Αυστρία. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα αυτή τη σύμβαση, ούτε και με το προαιρετικό πρωτόκολλο. Απλά και στις δύο περιπτώσεις λέμε ότι το Κοινοβούλιο εγκρίνει τα πορίσματα της σύμβασης, το περιεχόμενο μάλλον της σύμβασης και του πρωτοκόλλου. Έχουμε προετοιμάσει αυτό το σχέδιο ψηφίσματος λοιπόν. Ευχαριστώ τους συναντέλφους που έχουν υποβάλει τροπολογίες. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Απλά ε, για... υπάρχουν κάποιες τροπολογίες για ε, τις ένοπλες δυνάμεις της Ένωσης, τροπολογία 3 συγκεκριμένα. Έγραψα στους συναδέλφους που ε, συνέταξαν αυτή την τροπολογία και τους ζητώ να το ξανασκεφτούν. Μου έδωσαν διευκρινήσεις, βέβαια, Απλά λέμε, καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποσύρει την επιφύλαξή της. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ε, τροποποιηθεί η οδηγία ε, του 78 που συνιστά το γενικό πλαίσιο ούτως ώστε να γίνει συμβατή οδηγία με την σύμβαση αλλά ε, το να επαναδιαπραγματευτούμε αυτή την οδηγία 78 ε, και να την αναθεωρήσουμε θα ήταν αντιπαραγωγικό και θα ε, αναστείλει ή θα ανακόψει τελείως τη διαδικασία προσχώρησης και κύρωσης της σύμβασης και του πρωτοκόλου. Αυτό ήθελα λοιπόν να σας αναφέρω και Κλείνω την παρέμβασή μου λέγοντας, ευχαριστώντας και πάλι και τους συναδέλφους που έβαλαν τροπολογίες και τη γραμματεία που με βοήθησε πάρα πολύ στη σύνταξη του ψηφίσματος. Σας ευχαριστούμε κυρία Γέλεβα. Θα ήθελε κάποιος το λόγο. Κανείς δεν έχει ζητήσει το λόγο. Α, η κυρία Λίν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ γιατί εργαστήκατε σκληρά και συνεργαστήκαμε στενά. Υπήρξαν κάποιες δυσκολίες, γιατί αλλάξαμε κάπως τη στάση και τη γραμμή που... Κάποιος μου κάνει νοήματα, γι' αυτό σταμάτησα, Πρόεδρε. Είμαι σκιώδης ε, και έχω ασχοληθεί έντονα με το θέμα και... Και είναι πολύ καλή η γνωμοδότησή μας. Στην ε, οδηγία 78 υπάρχει μια εξαίρεση. Αν ε, προσπαθήσουμε να την αφαιρέσουμε θα χρειαστούμε πάρα πολύ χρόνο. Όχι ότι προτείνω να καταψηφίσουμε τροπολογία 3, όχι γιατί οπωσδήποτε είμαι κατά της άποψης αυτής, αλλά θεωρώ ότι είναι καλό να την υπερψηφίσουμε Υπάρχει ο κίνδυνος να καθυστερήσουμε λίγο τη διαδικασία. Απλά θα πρέπει να μεριμνήσουμε ούτως ώστε να κυρώσουν γρήγορα ε, όλα τα κράτη-μέλη της σύμβασης. Ε, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα με τις συμβάσεις του ΟΗΕ. Δεν υπάρχουν πολλοί που προσχωρούν. Για την κύρωση, για την προσχώρηση. Γι' αυτό θα πρέπει να αγωνιστούμε. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για τη δουλειά που κάνετε. Είναι πολύ καλή η γνωμοδότησή μας. Η Ρία Ομρόιτεν έχει ζητήσει το λόγο. Ε, ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω ως προς την έκθεση αυτή, αλλά θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι Στα τέλη της δεκαετίας 40, τα Ηνωμένα Έθνη κατάρτισαν μια χάρτα σε σχέση με την συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία. Μπορείτε να μου πείτε τι γίνεται με αυτή τη σύμβαση την 1748. Ποια ήταν η τύχη της. Δεν έχω ιδέα, λέει ο Πρόεδρος. Δεν ε, ζητά κανένας άλλος το λόγο. Ρίτσαρτ Χάουιτ. Ζητώ συγγνώμη διότι προσήλθα μετά από την ε, εισήγηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εργασία της και δεν μπορώ να αναφερθώ παρά στις ε, τροπολογίες ε, του υποφαινομένου και άλλων. Ως προς την τροπολογία 11 μιλάμε για μια εκστρατεία των κρατών μελών να προσυπογράψουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων το μας είχε απασχολήσει εξ αρχής, μιλώντας δηλαδή για τη σύνταξη μιας σύμβασης και είχαμε επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι όλα τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να επικυρώσουν καθώς και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ως θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει ο κίνδυνος να προσυπογραφεί και τα κράτη να πούνε «Α, τώρα αυτό έγινε, το θέμα θεωρείται λήξαν». Δεν θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Σε σχέση με την τροπολογία 13 και την οδηγία κατά των διακρίσεων, mainstreaming, εκπαίδευση. Αυτό είναι ένα διφορούμενο ζήτημα το οποίο όμως δεν θα πρέπει να βάλουμε κατά μέρος. Αυτό το αναφέρω εδώ και χρόνια, διότι άτομα με αναπηρίες θεωρούν ότι την χάνουν διακρίσεων και αυτό αφορά και παιδιά τα οποία θέλουν να συμμετέχουν στην κυρίως εκπαίδευση και δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και η επιλογή ε, αυτή δεν ε, χορηγείται προς τα παιδιά με αναπηρίες και εντάσσεται στην οδηγία κατά των διακρίσεων με βάση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό προσπαθώ να κάνω στην τροπολογία 11 ως προς την 15. Ε, και θα ήθελα και η Επιτροπή να απαντήσει για να είναι πραγματική, για να υλοποιηθεί δηλαδή η σύμβαση, θα πρέπει να έχουμε εφαρμόσει τις βασικές της αρχές. Και αυτό δεν αφορά την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης ή για τη Γενική Διεύθυνση που ασχολείται με αναπηρίες. Αφορά την εποπτεία ολόκληρης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μην αντιταχθούμε στη σύμβαση αυτή, να γίνουν οι κατάλληλες προσαρμογές. Ε, δεν μας απασχολούν μόνο θέματα αναπηρίας. Θα ήθελα όμως το υπεύθυνο τμήμα να αναφερθεί και σε αυτό, διότι θα πρέπει να ανταποκριθούμε έτσι ώστε να εφαρμόσουμε αυτές τις πολιτικές. Ως προς την οδηγία κατά των διακρίσεων και σε σχέση με την τροπολογία 16 αφορά την πλήρη εφαρμογή του ανεξάρτητου ρόλου των οργανώσεων που ασχολούνται με άτομα με θέματα αναπηρίας, αλλά και ανεξάρτητους οργανισμούς για την εφαρμογή της οδηγίας, για να την εξασφαλίσουν γιατί εδώ μιλάμε για την τήρηση των αρχών του Παρισιού και ήδη σε ορισμένα κράτη-μέλη ε, ισχύει κάτι τέτοιο και η Επιτροπή θα μπορούσε ίσως να μας δώσει μία απάντηση. Τάσομαι υπέρ της έκθεσης, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια και εδώ πιστεύω ότι θα υπάρξει μεγάλη ευρεία συνένεση και το ζήτημα είναι κεφαλαιόδους σημασίας γιατί έχουμε εργαστεί εδώ και χρόνια. Είναι ιστορική στιγμή ε, η στιγμή της συμφωνίας της σύμβασης και εμείς θα πρέπει να εφαρμόσουμε τις αρχές αυτές της σύμβασης για να αποτελέσουμε παράδειγμα για την Ήπειρό μας και τον υπόλοιπο κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν και το τελευταίο ομιλητή στον κατάλογό μου. Άρα η κυρία Γέλεβα μπορεί να συνοψίσει. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σημερίζομαι. τα περισσότερα από τα σχόλια των συναδέλφων και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους γιατί μας έκαναν πολύ καλές υποδείξεις και μιλήσαμε και για τη δέσμευσή μας ως προς τα άτομα με αναπηρία και τα σώμαστε και υπέρ της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών βεβαίως. Θεωρώ ότι η εφαρμογή της Σύμβασης και το προαιρετικό πρωτόκολλο των κρατών μελών για τα κράτη-μέλη που θέλουν να προσχωρήσουν είναι πολύ σημαντικό. Τώρα θα πρέπει να αποστείλουμε ένα μήνυμα από τη δική μας συζήτηση με την δική μας εργασία και ζητούμε και από τους άλλους να προσχωρήσουν το ταχύτερο δυνατόν. Ιδιαίτερα ως προς το προαιρετικό πρωτόκολλο που αφορά την εφαρμογή της σύμβασης σε σχέση με τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία. Χαίρομαι γιατί φτάσαμε σε ένα συμβασμό ως προς αυτό το κείμενο για να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να κινηθούν προς την ε, κύρωση της σύμβασης στο σύνολό της και να δεχτούν και το προαιρετικό πρωτόκολλο. Συμφωνώ. <coughs> τα, με τα σχόλια του κ. Χάουιτ και θα ήθελα να του πω ότι υποστηρίζουμε την τροπολογία του υπαριθμού 15. Νομίζω ότι στις προγενέστερες ε, συναντήσεις μας κατέστησα φέσο ότι τώρα θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην, ε, στην εργασία αυτή υπέρ της ε, οδηγίας του πρωτοκόλου και της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών έτσι ώστε να αποστείλουμε ένα σαφές μήνυμα χωρίς να περιλάβουμε άλλα θέματα στη συζήτησή μας. γιατί σε σχέση με την οδηγία του 78 είχε καθυστερήσει η κύρωσή της από τα κράτη-μέλη. Ελπίζω να φτάσουμε σε ευρεία συνένεση και μια πλειοψηφία, ευρεία πλειοψηφία έτσι ώστε να δείξουμε στα άτομα με αναπηρία ότι τασόμαστε υπέρ της σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σε ένα τόσο σημαντικό θέμα διότι εν των ευρωπαϊκών εκλογών Θέλουμε η Ευρώπη να βρεθεί πιο κοντά στους πολίτες, ιδιαίτερα αυτούς που έχουν υποφέρει πολύ στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται λοιπόν εδώ η συζήτηση των ε, σημείων αυτών για τη Συμβάση των Ηνωμένων Εθνών και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο. Η ψηφορία θα γίνει αύριο. Και τώρα... Έχουμε ακόμα δύο θέματα που έχουν συζητηθεί ήδη στο Συνδεσμό συστημάτων κοινωνική ασφαλεία τη διαδικασία εφαρμογή και το παράρτημα 11 για το οποίο είναι υπεύθυνο ο Γιάν Κρέμερ. Η κυρία Λάμερ πρώτη. Thank President. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Όπως ε, θα ξέρουν οι συνάδελφοι, ο εφαρμοστικός αυτός κανονισμός σχετίζεται με τον 8834 για τα συστήματα αυτά της κοινωνικής ασφάλισης και αναφερόμαστε στη δυνατότητα ηλεκτρονικής αναλύγης πληροφοριών πράγμα που ελπίζουμε ότι θα είναι πολύ πιο γλίγορο και πιο ακριβές από τη σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους και ηγητές, εκείνους που επέβαλαν τροπολογίες για τη συνεργασία τους. Γιατί αυτή τη στιγμή Εάν ψηφίσουμε αύριο υπέρ των συμβασικών τροπολογιών που έχουμε μπροστά μα θα είμαστε σε θέση να συμφωνήσουμε στη δεύτερη ανάγνωση με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ αυτούς που υπέβαλαν τις απολογίες και εκείνους που μπορούν έτσι να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο. όσον αφορά τις προσπολογίες αυτές, πετύχαμε κάτι σχετικά με τα χρονικά όρια. Όχι τόσο όσο θέλαμε, αλλά νομίζω αρκετά. Μπορούμε να έτσι να τελειοποιήσουμε το σύστημά μας. Όσον αφορά λοιπόν αυτά τα χρονικά όρια, έχουμε τώρα μια δέσμευση στις συμβαστικές τροπολογίες α και γ όσον αφορά το γεγονός ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν υπόψη τα δικά τους χρονικά όρια, δεν το έχουν κάνει μέχρι στιγμής, και τις συστάσεις που θα πρέπει να υπάρχουν χρονικά αυτά όρια μέσα σε κάποιες προθεσμίες ε, εντός των οποίων συγγνώμη, θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε αιτήσει ε, μεμονωμένων ατόμων ή οργάνων. Δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε περισσότερο αυτή τη στιγμή. Επίσης, <clears throat> έχουμε την τροπολογία 86, για στο άρθρο 86.1 που αφορά τον κανονισμό εφαρμογής και προβλέπεται μια συγκριτική αναθεώρηση για να δούμε κατά πόσο έχει βελτιωθεί αυτό το θέμα των χρονικών ορίων για την αλληλεγγύη πληροφοριών. Και έτσι, αν το δεχτεί το Σύμβουλο, θα ξέρουμε κατά πόσο τα πράγματα βελτιώνονται ή όχι. Όσον αφορά τους άμεσα ενδιαφερόμενους, το Κοινοβούλιο μας υπενθυμίζει ότι αυτό δεν αφορά μόνο την επικοινωνία μεταξύ ορισμικών οργανών, αλλά μεταξύ μεμονωμένων ατόμων. Στην εθνολογική σκέψη 21 έχουμε την τροπολογία 6 που αναφέρει τις διάφορες κατηγορίες. πρέπει να εξηγήσουμε τι εννοούμε δεν μπορούσαμε να έχουμε μία, ένα πλήρη ορισμό. Αλλά τώρα υπάρχει τουλάχιστον μία ένδειξη μέσα στα πλαίσια της εκλογής σκέψης 21. Στο άρθρο 3.1 προχωρήσαμε και έχουμε βάλει εδώ τώρα την υποχρέωση χορήγησης πληροφοριών. Είναι από τα ουσιαστικά θέματα που μας ενδιαφέρουν. Επίσης βρήκαμε μια λύση για το θέμα των πληροφοριών που δίνονται και είπαμε ότι θα πρέπει οι πληροφορίες αυτές να δίνονται γραπτά όσον αφορά την εφαρμοστέα νομοθεσία ως ισχύει μεταξύ των δύο χωρών, ιδίω στην περίπτωση ταπών εργαζομένων. Ε, είπαμε ότι αυτό θα πρέπει να ενταχθεί στο άρθρο 15.1 που αφορά αυτούς ακριβώς τους εργαζόμενου και νομίζουμε ότι αυτό είναι πολύ καλό. Σχετίζεται άμεσα με το πρόγραμμα που προσπάθησαν να λύσουν οι συνάδελφοι. Έχω πετάξει γλώσσα μου, δεν ξέρω τι λέω. Τέλος πάντων, ε, αυτά είναι τα προβλήματα που προσπαθούμε να λύσουμε είναι μικρό βήμα προς τα αλλά τουλάχιστον μας δίνει τη δυνατότητα να βοηθήσουμε τους ενδιαφερόμενους, όπως αναφέρεται σας είπα στο Επιλογή Σκέψη 21 και να τους δώσουμε κάποια ασφάλεια να ξέρουν τι γίνεται και να είμαστε σίγουροι ότι έχει δοθεί η ε, απαραίτητη ενημέρωση. κάποιες από τις ομάδες είπαν ότι προτίθεται να δεχθούν τις συμβαστικές ε, τροπολογίες που ε, προετοιμάσαμε και που μπορεί να δεχθεί και το Συμβούλιο. Και ότι αυτή θα είναι η θέση και της Επιτροπής μας και της Ολομέλειας όταν ψηφίσουμε επιτέλους μετά από όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γιάνν Κρέμερς. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εργαστήκαμε ε, εδώ ως διάδα. Άρα θα ήθελα να αναφερθώ σε εμάς και όχι σε μένα, πρώτο πρόσωπο πληθυντικού δηλαδή. Αυτά τα δύο θέματα, σε αυτά τα δύο θέματα δεν υπάρχει απόλυτη σύμπτωση απόψεων. Και για να είμαι πιο σαφής θα ήθελα να πω και με βάση που, αυτά που ε, προϋπόθηκαν αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ποιες τροπολογίες συμβασμού μπορούν να τύχουν συμφωνίας, διότι μας απασχολούσαν και θέματα σύνταξης διότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να διασαφίσουμε ορισμένα ζητήματα και στην πρώτη ανάγνωση είδαμε ότι το θέμα αυτό είναι ένα θέμα εκτέλεσης, εκτέλεσης από τις δημόσιες αρχές. Οι τροπολογίες είναι τροπολογίες ουσίες που μπορούν να αποσωφηνήσουν καλύτερα το κείμενο. Εν πάση περιπτώσει η δική μου ομάδα θέλει να προτείνει αυτό το κείμενο συμβασμού Λάμπερτ και τελευταίο θέμα σε σχέση με αυτή την έκθεση νομίζω ότι η αναβολή ή μάλλον για το πω διαφορετικά η αποστολή πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους εξαρτάται και από την ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών μεταξύ αρχών. Έτσι μπορούμε να φτάσουμε σε μία βελτίωση. Και ιδιαίτερα στο άρθρο 9 υπάρχει μία εγγενής ε, λογική. Εάν μεταφερθεί το άρθρο 9, από το άρθρο 9 στο άρθρο 15 αυτός ο ορισμός θα ήταν καλύτερα. Τώρα για να σχολιάσω τα δικά μου. Στην προηγούμενη συνεδρίαση είχαμε ανακοινώσει ότι φτάσαμε σε ορισμένους συμβιβασμούς που αναφέρονται στο παράρτημα 3, διότι υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη που κάνουν, ε, προβαίνουν σε μία εξαίρεση. Γιατί θα ήθελαν να αποσυρθούν από το παράρτημα. Άλλα κράτη-μέλη είπαν ότι θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτό το παράρτημα. Στη συνέχεια έγινε μία ζωηρή συζήτηση για τις επιπτώσεις αυτού του παραρτήματος υπαριθμών 3 και τέλος συμφωνήσαμε με την πενταετή αναθεώρηση, αλλά υπάρχει και ένας όρος για την αναθεώρηση αυτή. Δηλαδή να δούμε ποια θα ήταν η συνέχεια που θα δοθεί σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής, το κόστος, τη συχνότητα και ούτω καθεξής. Και τα περισσότερα κράτη-μέλη είπαν ότι θα πρέπει αυτή η αναθεώρηση να γίνει πριν λήξει η προθεσμία. Άρα ε, δεν έχουμε λόγο να μην εγκρίνουμε τον συμβιβασμό αυτό. Στην πρώτη σύνοδο μετά από αυτή τη βδομάδα μπορούμε να ψηφίσουμε νομίζω. Να το διεκπαιρεώσουμε το θέμα. Ε, Σας ευχαριστούμε. Δύο μιλήτες έχουμε. Η κυρία Στάουνερ και η κυρία Γιουκνεύνιτσνιέ. Θα είμαι σύντομη. Θέλω να σας ευχαριστήσω ένθερμα για τη συνεργασία μας και ζήτησα το λόγο απλά για να αναφέρω ότι ε, ήραμε τις επιφυλάξεις μας για τις συμβαστικές C και F, γάμα και σίγμα Μας είπε η εισηγήτρια ότι τα κράτη-μέλη που ακόμη δεν έχουν προθεσμίες ε, για τις ε, ανακοινώσεις ε, πρέπει να τις προσδιορίσουν. Μπορούμε να άρουμε τις επιφυλάξεις μας και στο όνομα της αρχής της επικουρικότητας καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Ευχαριστώ και υποστηρίζω πλήρως αυτή τη γνωμοδότηση. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Σας ευχαριστώ, κυρία Λάμπερτ. Ε, οργανώσατε με εκπληκτικό τρόπο τις εργασίες μας εδώ και τη συνεργασία σας με το, Κοινοβούλιο, με το Συμβούλιο συγγνώμη, και την Επιτροπή. Θα ήθελα να τονίσω αυτό που ανέφερε και η Τζιν Λάμπερτ, ότι δηλαδή η πολιτική μου ομάδα θα υποστηρίξει τις συμβαστικές τροπολογίες σας. Έχω ήδη στείλει γραπτό στην απάντησή μας. Υποστηρίζουμε λοιπόν τις ε, συμβαστικές ε, τροπολογίες. Υπενθυμίζω στους συναδέλφους δε ότι αυτή η γνωμοδότηση είναι πιο σημαντική όπως και άλλα έγγραφα που συζητήσαμε σήμερα, δηλαδή την ε, πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Η γνωμοδότηση αυτή φέρει επί της κοινωνικής προστασίας των πολιτών της Ένωσης και Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία σε εθνικές ορμοδιότητες, δηλαδή για την έγκαιρη κοινοποίηση ως προς τα κοινωνικά δικαιώματα από πλευράς του κράτους μέλους και δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στον συντονισμό των εθνικών συστημάτων. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε πόσο ε, μεγάλες ευθύνες καλούνται να επομιστούν τα κράτη-μέλη. θα είναι πολύ σημαντικές επιπτώσεις για τα κράτη-μέλη. Και άρα υποστηρίζω όλες τις προτάσεις ε, που συνηγορούν υπέρ της έκκλησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί ε, τις εθνικές δραστηριότητες ε, σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων που έχουν κέρια σημασία για τους πολίτες. Λοιπόν, συγχαίρω εκ νέου την κυρία Λάμπερτ και όταν τελικά εγκρίνουμε αυτό το τόσο σημαντικό έγγραφο θα, τελικά θα καταλάβουν οι πολίτες Ένωση ότι για αυτούς εργαζόμαστε εδώ στο Κοινοβούλιο. Ε, κυρία Ομερό ήταν. Ευχαριστώ. θα ήθελα να κάνω μία σύντομη παρατήρηση. Θυμάμαι ότι το 97-98 ε, μετήχα σε μία εκδήλωση ή μάλλον σε μία ε, συνεδρίαση για την ε, αναθεώρηση του κανονισμού 1408. Δέκα χρόνια διήρκησε η διαδικασία αναθεώρησης και πέρασε απαρατήρητη από η διαδικασία, αλλά για, εκατο... για πολλά εκατομμύρια πολίτες ο κανονισμός αυτός είχε πολύ πρακτικές επιπτώσεις στην καθημερινή του ζωή, οπότε πρέπει να γίνει μνήα. Ε, ήταν αξιόλογες προσπάθειες που έγιναν. Πολλοί συνάδελφοι συμμετείχανε, ε, μεταξύ των οποίων και Τζιν. Σε ευχαριστώ Τζιν, αλλά ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. και είναι οι θύνοντες ε, και οι συνάδελφοί σας που ήταν αρμόδιοι εκείνη την εποχή για αυτό το φάκελο εργάστηκαν με εξαιρετικό τρόπο και Ελπίζω να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα ε, στην προεκλογική μας εκστρατεία. Θέλει να προσθέσει τίποτα η συγγητρία. Τζιν. Ζαν, Τζιν. Ναι, Τζιν. Ναι, ε, θα είμαι σύντομη. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τα καλά τους λόγια. Είναι προϊόν συλλογική προσπάθειας αυτή η γνωμοδότηση. Θέλω να ευχαριστήσω τη γραμματεία, να μην το ξεχάσω, με βοήθησαν πάρα πολύ και ευχαριστώ και την Επιτροπή. Ανέλαβαν ε, σοβαρή δέσμευση, είχαν αυτή την πεποίθηση που χρειάζεται, ώστε να έχουμε ένα αποτέλεσμα ευνοϊκό για τους πολίτες τελικά μας βοήθησαν μετά από κάποιες δυσκολίες που είχαμε. Ελπίζω να μην συμβεί κάτι τραγικό μέχρι την αυριανή ψηφοφορία. Και μετά θα περάσουμε, θα περάσει η έκθεση και από την Ολομέλεια, όπου θα είμαι, ε, θα ακούσουν ε, τα φιλικά μου λόγια όλοι όσοι συνεργάστηκαν μαζί μου. Ναι, ναι, όλα καλά θα πάνε αύριο. Πήρα επιστολή από το Συμβούλιο, δε, ότι συμφωνούν το έχετε εδώ, άμα το θέλετε. Αύριο θα ψηφίσουμε. Ε, ολοκληρώνουμε και αυτό το σημείο. Το τελευταίο σημείο περνάμε τώρα. Δεν θα συνεδριάσουν οι συντονιστές γιατί συμφωνούμε με τις προτάσεις της γραμματείας. Το τελευταίο σημείο λοιπόν που θα συζητήσουμε σήμερα είναι η ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα. Ο κύριος Σίλβα Πινέντα. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για το ενδιαφέρον τους για αυτή την έκθεση. Έχουν υποβληθεί 200 τροπολογίες και η πλειοψηφία κινείται προς την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή μεγαλύτερη κοινωνική συνένεση από τις 22 τροπολογίες μου και που υπέβαλα με τον κύριο Εσκομπάρ προσπαθώ να αντικατοπτριστούν οι επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής κρίσης και κοινωνικής κρίσης που πλήττει την Ευρώπη και τον κόσμο. Εξετάστηκαν εκ του μαζί με την Επιτροπή Γυναικών και Ισότητας των Δύο Φύλων, μαζί με τις Επιτροπές ε, Περιβάλλοντος, δημόσια Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Οι συζητήσεις ήταν επικοδομητικές και μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα με 26 τροπολογίες συμβιβασμού και δύο προφορικές τροπολογίες. Αυτή η διαδικασία φτάνει σε μία ε, εξισορροπημένη έκθεση με βάση τις προτεραιότητες της κοινωνικής ατζέντα. Θα ήθελα να δούμε τις ε, τροπολογίες συμβιβασμού δείχνουν ότι υπάρχει μία συνένεση καθώς και εξυγχρονισμός της ατζέντα, ιδιαίτερα σε επίπεδο συντάξεων υγείας και μείωση των κοινωνικών δαπανών σε καιρούς κρίσης. Επίσης, τις διαρθρωτικές ε, ε, αλλαγές στα κράτη-μέλη. Η Επιτροπή πολιτισμού και αθλητισμού συνεισέφερε και η έκθεση ε, Τσίμερ μας βοήθησε σε σχέση με την καταπολέμηση της φτώχειας με μεγάλη πλειοψηφία. Οι τροπολογίες poderia ajudar, por exemplo, outra. Α ε, και 3 ε, σχετίζονται και με τις ε, δημογραφικές προκλήσεις. Το δημογραφικό αναφέρεται και στην 6. Το F μιλά για την συμφωνία μεταξύ ομάδων σε σχέση με την εγκατάλειψη του σχολείου ως προς τη συγκρισιμότητα και αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων είναι κάτι το οποίο είναι θεμελιώδες για την εσωτερική αγορά σε σχέση με το AIDS μιλάμε για την ενσωμάτωση των ανθρώπων όταν βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας για να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια. Το ΙΟΤΑ μιλά για την αλλαγή ενεργοποίησης κοινωνικών πολιτικών και απασχόλησης για να αντιμετωπίσουμε την παρούσα κρίση με την απασχόληση και την απασχολησιμότητα καθώς και την ενεργό συμμετοχή. Το J αναφέρεται και στην έκθεση τόγια που ε, ενέκρινε το σώμα με μεγάλη πλειοψηφία και αφορά την κοινωνική δράση. Το ΚΑΠΑ μιλάει για τις μικροπιστώσεις για την ένταξη των ανθρώπων στην αγορά εργασίας, δημιουργώντας δικές τους επιχειρήσεις. Η ΕΛ μιλάει για τις κοινωνικές διαδικασίες με βάση την επικορικότητα και τα, τα νέα μισθολογικά με την ε, μεγαλύτερη συμμετοχή των ανέργων. Το F αφορά τις ε, αρνητικές επιπτώσεις της μετανάστευσης στις χώρες υποδοχής, μάλλον προέλευσης και να μην ξεχνάμε ότι η κατάσταση είναι ε, ιδιαίτερα κακή και στις χώρες υποδοχής. Οι και οκτώ μιλάν για τα δικαιώματα των εργαζομένων και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ε, κρίση έλλειψης εμπιστοσύνης σε σχέση με την χρηματοοικονομική κρίση. Το P μιλάει για την ε, πρόσβαση στην εργασία, το Q αφορά τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές πολιτικές που είναι συμπληρωματικού χαρακτήρα. Ε, όμικρον και 7 αναφέρονται στην ε, παρούσα χρηματοπιστωτική κρίση σε σχέση με την ανεργία. Οι δύο αναφέρεται στις πιο ευάλωτες κατηγορίες σε σχέση με το κίνδυνο φτώχειας. Η τέσσερα αφορά την, ε, την αρχή ενσωμάτωσης που μπορούμε να ε, εντάξουμε στην έκθεση. Η 70 και 75 της Γκαρμπίδα Κρετού ασχολείται με τα ελάχιστα δικαιώματα των εργαζομένων. Ξέρω ότι υπάρχουν ε, προβλήματα τα οποία μπορούν να συζητηθούν αύριο σε σχέση με θέματα λεπτομερίας και θα ήθελα να πω ότι στα πλαίσια της ε, κρίσης αυτής θα πρέπει να αναφέρουμε σαφώς ότι η Ευρώπη και οι κοινωνικές πολιτικές θα πρέπει να είναι πιο ενισχυμένες και αυτό, αυτός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της έκθεσης ε, σε σχέση με την κοινωνική ειρήνη που προσπαθούμε να επιτύχουμε. Ευχαριστώ τρεις ομιλητές, ε, Κρέμες, Κρετή και Λεγκέρ. Κύριε Κρέμες, <coughs> όχι, Κρετή. Ωραία, εσείς πρώτα. Θα ήθελα να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή που περιέγραψε την διαδικασία των διαπραγματεύσεων, αλλά όχι το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε όλες τις συμβαστικές τροπολογίες για τα έγγραφα αναφορά, τις παραθέσεις που γίνονται. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτό. Ε, Παρ' όλα αυτά θα κάνουμε κάποια σχόλια για τα εκτιμώντας τις ιδεολογικές σκέψεις μάλλον την αιτιολογία εννοεί η ομιλήτρια των συμβαστικών τροπολογιών. Δεν πρόκειται για ε, προϊόν συμβιβασμού ανάμεσα στις διάφορες πολιτικές ομάδες. Είναι κάποιες ενοποιημένες ε, τροπολογίες, ε, συγχωνευμένες τροπολογίες. Κάποιες πολιτικές ομάδες φάσουν να τις υποστηρίξουν απλώς. Και ζητώ από τον εισηγητή, διότι αυτό το θέμα έχει μεγάλη σημασία για μας. Να τον ρωτήσω λοιπόν, γιατί το ΕΛΚ δεν υποστηρίζει τροπολογία 46, που ζητά τη ρίση της ε, κειμένης εθνικής νομοθεσίας και του υφισταμένου πλαισίου. Μία τροπολογία που ζητά την τήρηση της ένομης τάξης δεν μπορεί να απορρίπτεται. Αφήστε που πρόκειται για τροπολογία για την αιτιολογική σκέψη. Δεν είναι μία δήλωση μέσα στο, διατακτικό μέσα στο κυρίως τμήμα του κειμένου. Ευχαριστώ που συμφωνήσατε για την τροπολογία 70 και 75 τελικά και τη σχέση ανάμεσα στις οικονομικές ελευθερίες και τα κοινωνικά δικαιώματα. Σας ευχαριστούμε, αλλά εμένουμε στη θέση μας για τις τροπολογίες 65 έως και 68. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε σε συμβασμό, αλλά Ανάμεσα στους σοσιαλιστές και τον εισηγητή υπάρχει χάσμα. Ε, μεγάλη διάσταση απόψεων. Εμείς απευθύνουμε πολύ περισσότερες επικρίσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ το ΕΛΚ είναι πολύ πιο ικανοποιημένο με την ε, ένομη τάξη, με, την, ε, με το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει. Υπάρχουν κάποιοι τομείς όπου ε, χρειάζεται μία νομοθετική ρύθμιση. Για τις ε, τροπολογίες που σχετίζονται με το ίδιο το περιεχόμενο, έχουμε ε, μία επιφύλαξη για την τροπολογία L. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε και δεν θα την υποστηρίξουμε, λοιπόν. Μπορούμε να υποστηρίξουμε τις λοιπές τροπολογίες που προτείνει ο εισηγητής. Αλλά διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας για αυτά που προανέφερα και ο Γιάννη υποθέτω θα ε, συμφωνήσει μαζί μου, θα πάρει το λόγο τώρα. Ο κύριος Κρέμες και ο κύριος Λέιντε ακολουθούν. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομο ε, γιατί θα είπε η μου, η κυρία Κρετή αυτά που ήθελα να αναφέρω. Απλά επανέρχομαι στο... στην ενδυνά... στις ενδεχόμενες επιπτώσεις αυτού του... αυτής απόφασης. Ε, τον Ιούλιο πέρσι ε, εξεδόθη η αναθεωρημένη, ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ειδικά στη δική μας πολιτική ομάδα απευθύναμε πάρα πολλές επικρίσεις διότι η πρόταση της Επιτροπής όχι μόνο ήταν περιορισμένου εύρους αλλά έφτασε και αργοπορημένη. Δεν πρέπει να κάνουμε λοιπόν το ίδιο λάθος αυτή τη φορά. Χρειαζόμαστε μια πολύ πιο φιλόδοξη κοινωνική ατζέντα. Γι' αυτό και υποβάλαμε τόσες πολλές τροπολογίες που δίνουν ε, λίγη περισσότερη ουσία ε, στο κείμενο. Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε τις προθέσεις της σοσιαλιστικής ομάδας. Θέλουμε οι κοινοτικές, οι ευρωπαϊκές δραστηριότητες να συνδεθούν με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Ε, ε, κάναμε μια επίσκεψη και υπέβαλα τη σχετική έκθεση. Σε παγκόσμιο επίπεδο θα έπρεπε να είναι δυνατόν να ε, καταλήξουμε σε συμβάσεις σε τριμερές επίπεδο, δηλαδή να εκπροσωπούνται οι εργαζόμενοι εργοδότες και οι κυβερνήσεις, όπως στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Αυτό θα μπορούσε να ήταν το εφαλτήριο για να δρομολογηθεί ένα πολύ πιο φιλόδοξο πρόγραμμα. Αυτό το πνεύμα διαπνέει πολλές από τις τροπολογίες μας ε, και κάτι άλλο που μάλλον θα είναι δύσκολο να συζητηθεί σήμερα εδώ στην Ευρώπη, βιώσαμε κάποιες εξελίξεις στον κοινωνικό τομέα για την κοινωνική ε, πολιτική είχαμε τα σλόγγαν ε, ενότητα και διαφορετικότητα. Τι σημαίνει αυτό ότι πρέπει να τηρείται το υφιστάμενο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο που βασίζεται σε δύο βασικά συλλογικά όργανα, δηλαδή εργατικό δίκαιο και συλλογικής διαπραγματεύσεις. Αυτά είναι τα δύο σκέλη. Και τα τελευταία χρόνια είδαμε ότι αυτή η ενότητα και η διαφορετικότητα που έπρεπε να αποτελέσουν το έρισμα της κοινωνικής πολιτικής τελικά μετεξελίχθηκαν σε μια διεθνική προσέγγιση από πλευράς και Επιτροπής και ΔΕΚ. Και θεωρούμε ότι είναι πολύ περίεργο που σημειώθηκαν αυτές οι εξελίξεις χωρίς να γίνει ουσιαστικά πολιτική συζήτηση. Και φαίνεται και αυτό σε κάποιες από τις τροπολογίες μας. Είναι μια ανησυχία που έχουμε και πρέπει να γίνει η απαιτούμενη συζήτηση. Δηλαδή ποιος είναι αρμόδιος για τα κοινωνικά και οικονομικά αυτά ζητήματα στα κράτη-μέλη. Προσπαθούμε να, μέσα από τις τροπολογίες να συνδέσουμε το έγγραφο με κάποια θέματα της ε, πράσινης βίβλου της Επιτροπής, ε, γιατί δεν υπήρξε παρακολούθηση, δεν είναι δόθη συνέχεια. Ε, απευθύνουμε έκκληση στην Επιτροπή μέσα από τις τροπολογίες μας να δώσει συνέχεια σε αυτή τη βίβλο γιατί υπάρχουν ε, για το εργατικό δίκαιο πολλά σημαντικά στοιχεία μέσα στην πράσινη βίβλο που πρέπει να επεξεργαστούμε και αναπτύξουμε στο μέλλον. Με τελικό απότερο στόχο το Κοινοβούλιο να εκδώσει μια πιο φιλόδοξη έκθεση, δηλαδή να τονίζουμε ότι υπολείπεται πολύ σοβαρό έργο σε αυτόν τον τομέα. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Λεϊντέ και ο κύριος Κούστασε μετά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα, Πρόεδρε, καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έργο που επιτέλεσε και την ατμόσφαιρα στο οποίο έγινε αυτό. Η ατμόσφαιρα ήταν πάρα πολύ θετική. Ε, κάτι που κατανόησαμε πολύ καλά. Δεύτερον, υπάρχει ένα νέο στοιχείο βρίσκομαστε τις παραμονές της δεύτερης κορυφής αρχές Μαΐου και θα πρέπει νομίζω η Επιτροπή μας να σκεφτεί το εξή. Βέβαια, μπορώ να συμφωνήσω ότι υπάρχουν κάποια σημεία πάνω στα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε συζητήσει. Από την άλλη μεριά, νομίζω ότι έχουμε κάθε συμφέρον η δική μας Επιτροπή όσον αφορά τα θέματα πάνω στα οποία εργάζεται εδώ και πολύ καιρό να αποστέλει πολύ σαφή μηνύματα. Θα πρέπει να σκεφτούμε, να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην προσπαθούμε δηλαδή να υπερφωνοφτώσουμε το κείμενο. Το έγγραφο του κ. Σίλβα είναι πολύ σαφές, με σύνομες ε, παραγράφους, ακριβείς παραγράφους. Δεν επιτρέπεται λοιπόν να το υπερφωτρώσουμε γιατί αυτό θα αποδυναμώσει το μήνυμά μας. Χαίρομαι που μπορέσαμε να συμφωνήσουμε με τον εισηγητή και ελπίζω αύριο με το σύνολο της Επιτροπής όσον αφορά κάποιες τροπολογίες για τις ε, γενικές υπηρεσίες ε, γενικού συμφέροντος. Είναι ορισμένα πράγματα που τα έχει πάρει υπόψη το εισηγητής άμα μπορούμε να συμφωνήσουμε πάνω σε συμβαστικέ τροπολογίε και σε τροπολογίες τροπολογίε που ε, τη χάνουν υποστήριξη του εισηγητή, θα είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Κύριο Κουστάσοφ, σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ συμφωνώ με τι ευχαριστίε ε, και τα συγχαρητήρια για τον κύριο you όσον αφορά τις τροπολογίες του και όσον αφορά τις ε, συμβαστικές τροπολογίες που υπέβαλε και τις προσπάθειες που κατέβαλε για να συμφωνήσουν πάνω σε αυτό και σκιώδεις ηγητές. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Η φτώχεια είναι ντροπή, όχι για τους φτωχούς, για εμάς τους πολιτικούς, που δεν μπορούμε να την καταπολεμήσουμε τη φτώχεια. Καμιά φορά νομίζουμε ότι εάν δώσουμε σε όλους εργασία και προωθήσουμε την παραγωγικότητα θα έχουμε λύσει το πρόβλημα. Γι' αυτό και εγώ στην τροπολογία 17 αναφέρω συγκεκριμένα το ότι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές στατιστικές το 8% των εργαζομένων απειλούνται από φτώχεια. Δηλαδή η εργασία δεν προστατεύει απαραίτητα από την ένδια. Ε, θα ήθελα εδώ να αφαιρθώ και σε αυτά που είπε ο κύριο Κρέμερ, δηλαδή ότι η κοινωνική πολιτική δεν είναι και τόσο φιλόδοξη όσο θα έπρεπε. Πολλά θα πρέπει να γίνουν ακόμα. Ακόμα και αν απαριθμέται ποιο απειλείται από φτώχεια, δεν αναφέρονται οι μετανάστες, ιδίως οι μετανάστες που δεν έχουν χαρτιά, επίσημα έγγραφα. Βλέπουμε τι γίνεται στη Νότια Ιταλία, στην Αλμερία, στη Νότια Ισπανία, πώς μεταχειρίζονται εκεί τους ανθρώπους. Είναι πραγματικά ντροπή για την Ευρώπη που είναι δυνατόν κάτι τέτοιο να υπάρχει στην Ευρώπη. Ε, πρόσφατα σε ένα βιβλίο που μου χαρίσα διάβασα ότι 500.000 άνθρωποι, κυρίως γυναίκες, κυρίως γυναίκες που εργάζονται στην βιομηχανία του σεξ υποχρεωτικά, καταναγκαστικά, έρχονται κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Αυτά είναι τα στοιχεία που πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Με το πλούτο που έχουμε θα πρέπει να εγγυηθούμε όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς και με ελευθερία. Αυτό είναι δυνατόν μόνο εάν σκεφτούμε επιτέλους ότι θα δώσουμε ένα ελάχιστο εισόδημα σε όλους. Δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό. Δεν πρέπει να νομίζουμε ότι αυτό το πετύχουμε με πλήρη απασχόληση. Ουτοπία είναι αυτό. Θα πρέπει να κάνουμε μια ανακατανομή του εισοδήματος με πιο δίκαια φορολογικά συστήματα γιατί ξέρουμε ότι οι πραγματικά πλούσιοι, εκείνοι που έχουν τα μεγάλα κέρδη, δεν πληρώνουν φόρους. Πολλά πρέπει να γίνουν εδώ. Λοιπόν, εδώ θα τελειώσω ευχαριστώντας για άλλη μια φορά τον κύριο Σίλβα Πενέντα. Αλλά πραγματικά κύριε Κρέμερ, εμείς δεν κάνουμε αρκετά για τα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής. Πρέπει να κάνουμε παραπάνω. Ευχαριστώ, δεν έχει ζητήσει κάποιο άλλο το λόγο, οπότε θα δώσω το λόγο στον κύριο Σίλβα Πενέντα για να συνοψίσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο γενικής εμβέλειας. Ήθελα να είναι ένα σύντομο αυτό το κείμενο που να εστιάσει την προσοχή στα ουσιώδη ζητήματα. Δεν έχω τίποτα εναντίον των προτάσεων που έγιναν, ξεκινώντας από την κυρία Κρετού. Αλλά ε, ε, εάν προσθέτουμε, προσθέσουμε, θα χανόμαστε στο τέλος. Εντάξει, αν το θέλετε. Ο κύριος Κρέμερ ε, μίλησε για το Διεθνές Γραφείο Εργασίας έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει περισσότερα για να βοηθήσει το Διεθνές Γραφείο Εργασίας για την αξιοπρεπή εργασία με βάση τις ε, προδιαγραφές του ΔΟΕ έτσι ώστε να συνεισφέρουμε στην παγκόσμια ειρήνη και στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά τώρα θέλω να προσθέσει και κάτι άλλο που είναι ταυτόσιμο. Δεν υπάρχει τίποτα το διαφορετικό. Δηλαδή 162 λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσπαθήσει να επηρεάσει τους διεθνούς οργανισμούς για ε, αξιοπρεπή εργασία, ιδιαίτερα με βάση τις συμβάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Εγώ δεν έχω τίποτα εναντίον. Αλλά στο τέλος τι θα κάνουμε. Θα είμαστε επαναληπτικοί, δηλαδή θα χανόμαστε ως προς την ουσία σε σχέση με τις προτεραιότητές μας Άρα δεν ε, έχω τίποτα εναντίον των ε, τροπολογιών, αλλά θεωρώ, όπως ήδη είπε κάποιος, ότι βάζουμε περισσότερα στο λίδια, στο χριστουγεννιάτικο δέντρο και στο τέλος όλα είναι θέματα προτεραιότητας. Αλλά δεν έχω τίποτα εναντίον της συμπερίληψης ορισμένων ε, τροπολογιών ως προς το περιεχόμενο, ως προς τον ε, τύπο, εν πάση περιπτώσει. Αν ε, το κρίνετε ότι συμβαδίζει τύπος με περιεχόμενο, μπορούμε να, το, μπορούμε να κάνουμε μία αναθεώρηση, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχουν πολιτικά προβλήματα ουσίας. Νομίζω ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αποστείλει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα σε τρία-τέσσερα επιμέρους σημεία. Θα ήθελα να πω με την, προς τη σοσιαλιστική ομάδα ότι δέχομαι αυτά που είπατε, αλλά αυτά θα πρέπει να συσχετιστούν με τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και με την χρηματοπιστωτική κρίση. Αλλά η κοινωνική πολιτική υποχρησιμοποιείται αλλά πιστεύω ότι η Ευρώπη χρειάζεται μία πολύ μεγαλύτερη κοινωνική πολιτική. Πρέπει να την ενδυναμώσουμε. Εάν όμως προσθέτουμε, προσθέτουμε, προσθέτουμε, τότε διαχέεται το περιεχόμενο. Θα πρέπει η κοινωνική πολιτική να ενισχυθεί, να είναι το επίκεντρο με όλα τα μέτρα, με όλα τα μέσα. Αν δούμε ποιο είναι το πιο σημαντικό μέσο, τότε θα χαθούμε. Θα χαθούμε στη λεπτομέρεια αλλά άμα θέλετε μπορώ να το δεχτώ. Δηλαδή σήμερα ή αύριο το πρωί να δούμε το ένα ή το άλλο σημείο, αλλά ας μην κάνουμε κατάχρηση έτσι ώστε να μην έχει πολύ διασταλτικό περιεχόμενο και να μην βοηθάει σε τίποτα, να χάσουμε την ουσία δηλαδή. Er- Ευχαριστώ. Ήταν το τελευταίο σημείο. Κανείς δεν έχει εγγραφεί στον κατάλογο μιλητών. Να σας πω ότι αύριο θα ψηφίσουμε για αυτή την έκθεση. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την ενδιαφέρον σας. Αύριο στις 9 θα αρχίσουμε. Ο Πρόεδρος ευγενικά ευχαριστεί και τους διερμηνείς. Τον ευχαριστούμε και εμείς. Καλό βράδυ.